Good afternoon everybody and now let's continue with... Γεια σας λέει πρόεδρος. Ας συνεχίσουμε με την κυρίως συνεδρία της Επιτροπής. Πρώτα πρώτα να σας ε, πω, πληροφορίζω ότι έγινε συνάντηση των ε, συντονιστών το τέλος πριν από μισή ώρα πρώτα πρώτα εγκρίθηκε η μέρες για 21 και 22 Ιανουαρίου και 10 και 11 Ιουλίου. Αυτέ οι μέρε διατάξεις επομένως εγκρίθηκαν. επίση. και κάποιε αναφορέ για προστασία πτηνών, για το νέο φόρο ε, στις Βαλαιαρίδες, πάμε να πάνε τον Ιούλιο, το ζήτησε το ΕΛΚ και το EFTD. Και είπαμε να προσθεθούν και πιστές αναφορές ε, για τη συνάντηση του Σεπτεμβρίου και επίση είπαμε και για την απασχόληση των ε, αναπήρων επίσης όσον αφορά τις επίμαχες ε, συστάσεις και εκεί έκανα κάποια πρόταση γιατί μου είπαν ότι θα πρέπει να διαβάσουμε τους ε, ρυθμούς. Α, ξέρω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ε, βαρετό, αλλά πρέπει να γίνει αυτό για να είναι έγκυρη η αναφορά μας. Οπότε είπαμε 41-63, 15-14, ό,τι είπα εγκρίθηκε. Επίσης, όσον πρώτο 14-84, είπαμε να υπενθυμίσουμε ε, αυτά που πρέπει να κάνουν οι ρουμανικές αρχές τώρα όσον αφορά τα θέματα β' Κλείσαμε τις αναφορές 517, 1666, 652 και 733 και άλλες θα μείνουν ανοιχτές και θα γίνει επίσης ε, η σωστή παρακολούθηση των εξελίξεων όσον αφορά τώρα τις ακροάσεις ε, εγκρίθηκε η αποστολή στην ε, Ιταλία, στο Ταράντο, επίσης και το πρόγραμμα για την Λάρνακα στην Κύπρο, τη σχετική αποστολή δηλαδή, και όσον αφορά τη σύνθεση των αποστολών, τώρα όσον αφορά τους συντονιστές, άλλο εγκρίναμε τα της 22 Δευτέρου Ιουνίου για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνη των πολιτών για το Ευρωπαϊκό Όραμα, γραπτή διαδικασία και προσωρινό πρόγραμμα όσον αφορά την ακρόση για τους ενθογενείς. Επίσης είπαμε για την αναφορά 747 που αφορά τους ενθογενείς στις βαλτικές χώρες και αποφάσισαν το εξή οι συντονιστέ. Μου έδωσαν εντολή, ούτω ώστε να εμείνω για να περιληφθεί αυτή η αναφορά στην αυριανή συνάντηση με τον πρόεδρο τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Τώρα, όσον αφορά την παρακολούθηση των ελευθεριών για τον Brexit, είπαμε να υποβάλουν προτάσει οι συντονιστέ και να έχουμε ε, ένα ψήφισμα για τα βιώματα των πολιτών θα πάει στην ε, συνδυασία των Προέδρων και επίσης ε, μέχρι τέλος Αυγούστου με γραπτή διαδικασία να εγκριθεί αυτή η πρόταση. Επίσης όσον αφορά την ισότητα των φίλων για το πρόγραμμα δράσης μας, για το mainstreaming, ε, ο κύριος Γιάρ, ο οποίος το έχει αναλάβει, παρουσίασε ένα σχέδιο κειμένου για αυτό το πρόγραμμα δράσης που βάζουν οι συντονιστές να το εγκρίνουν στην επόμενη συνάντηση και επίσης να προτείνουν κάποιες τροπολογίες μέχρι τις 6 Ιουνίου. Οι συντονιστές ε, επίσης ενημερώθηκαν για την εκδήλωση του 10 Οκτωβρίου για τους αναπήρους και οι σοσιαλδημοκράτες ήδη έκανα κάποια πρόταση όσον αφορά το σχετικό εργαστήριο και που είπαμε ότι όποιος θέλει μπορεί να προβάλλει όποιο κομμάτι θέλει να προβάλλει προτάσεις. Επίσης αποφάσισαν οι συντονιστές να ζητηθεί από το Policy Department ε, ε, γάμα να μας ετοιμάσει ένα σχετικό κείμενο και να ενημερωθούν οι μελέτες οι οποίες ε, έχουν ε, προκύψει. Αυτά όσον αφορά τους συντονιστές και πρέπει να σας πω ότι ήμασταν στη συνάντηση των συντονιστών πάρα πολύ αποτελεσματικοί. Τόσο πολύ που είχαμε και χρόνο για ένα καφεδάκι πριν να αρχίσει η τωρινή συνεδρίαση. Άρα συγχαρείτε μας. Τώρα, εάν δεν υπάρχει κάποια ένσταση όσον αφορά την ημερήσια διάταξη, να την εγκρίνουμε. Θα ήθελα όμως να μετακινηθεί η αναφορά, η, το θέμα για την Ισπανία να πάει πριν την, ε, το, το σημείο που φορά την διαμεσολαβήτρια, αν συμφωνείτε. Τώρα θα εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης του Απριλίου 24 και 25 έχετε λάβει τα πρακτικά, δεν υπάρχει κάποια ένσταση τότε θεωρώ ότι τα εγκρίνεται. Δεν μου έχουν ζητήσει κάτι άλλο για τα διάφορα. Οπότε συνεχίζουμε και πάμε στην ψηφοφορία. Α, το Φεβρουάριο θα είμαστε στην Σουηδία. Δεν είναι το πιο ε, ιδιώδες από πλευράς καιρού, αλλά έχουμε αυτήν την επίσκεψη την οποία την κάναμε τότε πρέπει να ψηφίσουμε για το σχετική σύσταση και θα πρέπει να γίνει η ψηφοφορία. Amendment 1, who is in favor? Against? Abstentions? Approved. Amendment 2, in favor? Against? Τροπολογία 1, 2, εγκρίθηκαν οι 1 και οι 2, 3, υπερ κατά, αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 4 τώρα η ψηφοφορία κάτι σοβαρό 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και η οριστική ψηφοφορία δια της ηλεκτρονικής οδού άρχεται η ψηφοφορία υπέρ το οποίο σημαίνει πως μπορεί να κλείσει η ψηφοφορία το οποίο σημαίνει για να δούμε δεν είδα τους αριθμούς. 19.00, το οποίο σημαίνει 20.00. Μπράβο μας. Οπότε ας συνεχίσουμε με την παρουσίαση από την διαμεσολαβήτρια για το, είναι η ετήσια έκθεση για το έτος 2016. Η κυρία Ολοράιλη βρίσκεται καθοδόν Εντάξει, ας καλωσορίσουμε τώρα την διαμεσολαβήτριά μας, την κυρία Ορέιλη, η οποία θα μας παρουσιάσει την ετήσια έκθεση για το 2016. Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ μαζί μας και ανυπομονούμε για τα ευρήματά σας. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, καλό απόγευμα σε όλους. Χαίρομαι όπως πάντα πολύ που βρίσκομαι εδώ για να αναφέρω στην Επιτροπή αυτή και την εργασία του γραφείου μου κατά ε, το έτος 2016. Οπότε θα περάσουμε σύντομα κάποιες διαφάνειες με λεπτομερείς πληροφορίες ή μάλλον με τα κορυφαία σημεία της εργασίας μας. Μετά μπορούμε να ασχοληθούμε με ερωτήσεις. Η πρώτη διαφάνεια, βλέπουμε δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερα κάθε χρόνο. Πρόκειται για έρευνες που έγιναν το 2016 σε σχέση με τους ακόλουθους θεσμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για προφανείς λόγους είναι το μεγαλύτερο θεσμικό όργανο κατά του οποίου γίνονται καταγγελίες. Φυσικά έχει πάρα πολλή επικοινωνία με τους πολίτες τους ίδιους, με την πολιτεία των κινητών, με των πολιτών με επιχειρήσεις κτλ. Μετά έχουμε τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη δεύτερη θέση, στην τρίτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι βέβαια σε σχέση με την πολιτική του, αλλά με τη διαχείριση, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού, και έχουμε πολλούς υποψήφιους για μια θέση που έχουν αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα παραδείγματο χάρη δεν περνούν κάποιε εξετάσει ή αντιμετωπίζουν κάποιο άλλο πρόβλημα, οπότε απευθύνονται σε εμά. Για το Όλαφ επίση υπήρξαν ε, κάποιες καταγγελίες επίσης για άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμού. Όσον αφορά το αντικείμενο, το μεγαλύτερο ποσοστό αναφέρεται στην πρόσβαση σε έγγραφα 28% είναι ζητήματα προσωπικού αλλά δεν αφορά μόνο το προσωπικό εντός των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών αλλά έχουμε μια ιδιαίτερη νοοτροπία δυσκολία σε σχέση με την έψο καταγγελίες για σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με κάποιον ο οποίος σταματάει την εργασία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε μόνιμα είτε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα πηγαίνει στον ιδιωτικό τομέα, τότε υπάρχουν ανησυχίες κατά πόσον θα υπάρξουν συγκρούσεις συμφερόντων όταν από τον ιδιωτικό τομέα εισέρχονται οι υπαλλήλοι στην διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25% για την νοοτροπία παροχής υπηρεσιών έχουμε πολλές καταγγελίες πολιτών οι οποίοι μας λένε πως πολλές ε, ιστοσελίδες δεν έχουν μεταφραστεί στη γλώσσα τους Έχουμε καθυστερήσει στην επικοινωνία με τις υπηρεσίες. 18% των ερευνών <coughs> αποτελούν διαδικασίες επί παραβάση και την χρήση της διακριτικής ευχέρειας. Εμείς δεν έχουμε ενεργό ρόλο εκεί. Αυτό είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμείς απλά κοιτούμε αν όλες οι διαδικασίες εφαρμόστηκαν σωστά από την, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 14% των ερευνών αφορούν προκηρύξεις, συμβάσεις και επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές φορές υπάρχουν κάποιες διαφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάποιων και κάποιου άλλου συμμετέχοντα σε σχέση με κάποιο συμβόλαιο. Παραδείγματο χάρη όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πω ο ε, αντισυμβαλόμενο παρεύει κατά τη διάταξη, μια διάταξη του συμβολέου. Και 4% των ερευνών αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Παραδείγματο χάρη από την Frontex, τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά επίσης ε, εμπορικές συμφωνίε με χώρε όπω το Βιετνάμ. Και εξετάσαμε επίσης τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας σε σχέση με τους πρόσφυγες και τους ετούντες άσυλο, την οποία γνωρίζετε πολύ καλά. Αυτά, αυτές ήταν οι κύριες εκδηλώσεις, τα κύρια συμβάντα το 2016, τον Ιανουάριο. Απεσταλεί μια αποστολή σε μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών για να τους ευαισθητοποιήσουμε για τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεχάστηκαν για τη βοήθεια ανθρώπων είναι πόροι από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευση και Ένταξη. Υπήρξαν άνθρωποι που, παρα... που καταγγέλαν πω δεν ήξεραν πού βρίσκονται τα λεφτά, ποιο παρακολουθεί τη διαδικασία. Και το ζήτημα... για το ζήτημα αυτό απευθυνθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο. Τον Φεβρουάριο Απευθυνθήκαμε στην Επιτροπή, ζητήσαμε από την Επιτροπή να μας αναφέρει σχετικά με την άδεια κυκλοφορίας φυτοφαρμάκων, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι έρχονται στην, κυκλοφορία, στην αγορά χωρίς κίνδυνο. Τον, τον Μάρτιο σε σχέση, είχαμε μια έρευνα σε σχέση με την συνθήκη Ευρατών, Πρόκειψε ένα ζήτημα κατά πόσον κάποια βιογραφικά θα δημοσιευθούν ή όχι. Τον Απρίλιο η βελτίωση της διαφάνειας στο λόμπι του καπνού είχαμε μια εκδήλωση Τον Μάιο ανοίξαμε μία έρευνα για την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύγκρουση συμφερόντων ειδικών συμβούλων. Όπως γνωρίζετε κάθε επίτροπος έχει έναν ή δύο ειδικού συμβούλους. Έχουμε πάλι το ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων. Προσπαθούμε λοιπόν να διασφαλίσουμε πως δεν εμπλέκονται εξωτερικά συμφέροντα στην εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον Ιούλιο είχαμε διαφάνεια, το ζήτημα της διαφάνειας, τους τριμερείς διαλόγους. Απευθυνθήκαμε στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το θέμα. Είχαν θετική στάση επειδή όλοι περιμένουν μία απόφαση από το δικαστήριο σε σχέση με τη δημοσιοποίηση το διάσημο έγγραφο των τεσσάρων πυλώνων σε σχέση με τη διαμεσολάβηση και τους συμβασμούς που έγιναν και εκεί θα δείτε και οι ίδιοι Όπω υπήρξαν και άλλα ζητήματα με τα οποία ασχοληθήκαμε, τον Νοέμβριο παραδείγματο χάρη καλωσορίσαμε, επικροτήσαμε την δράση του Πρόεδρου Γιούνκερ για τον κώδικα δεντολογίας επιτρόπων. Το Δεκέμβριο είχαμε την Παγκόσμια Σύνοδο της εταιρική Σχέσης Ανοιχτής Διακυβέρνησης. Είχαμε το θέμα των, ε, το επίκαιρο θέμα των εναλλακτικών στοιχείων θα ήθελα να σας δώσω κάποια παραδείγματα επίσης. Κατά γελιών ρουτίνας που δεχόμαστε είναι η γλωσσική πολιτική για τη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπήρξαν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες οι διαβουλεύσεις γίνονταν μόνο στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά ενώ οι σελίδες της διαβούλευσης μεταφράζονταν σε όλες τις Ευρωπαϊκές Ένωσης και αυτό συνάδει με, δεν συνάδει με τις γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να φέρει τους πολίτες πιο κοντά όσον αφορά την ε, προσβασιμότητα των, ε, των δημόσιων διαβουλεύσεων. Εκεί υπάρχει ένα δημοκρατικό έλλειμμα, τώρα θα μεταφραστούν τα κείμενα αυτά σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο, η δεύτερη κουκίδα εκεί αναφέρεται σε επιχορηγήσεις και συμβόλαια. Έχουμε ένα πολωνικό Ινστιτούτο το οποίο έλαβε υπεργολαβικά μια εργασία. Η Ευρωπαϊκή Θεώρηση ε, Επιτροπή θεώρησε πως δεν είχε το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Ζήτησε 86.000 86 ε, ευρώ πίσω. Ήταν ένα τεράστιο ποσό. Ζητήθηκε μέσω email Είχαμε κα, καθυστερήσεις για καταγγελίες παράβασης. Λοιπόν, το 90% της εργασίας που διεκπερώνουμε σχετίζεται με μεμονωμένες καταγγελίες. Μίλησα για τη στρατηγική εργασία που κάνουμε, αν δούμε κάτι για το οποίο πιστεύουμε πως με μία μόνη έρευνα μπορούμε να ασχοληθούμε με πολλαπλά ζητήματα, τότε πιστεύουμε πως αυτό προσδίδει προστιθέμενη αξία στο ζήτημα, θα, θα επιλέξουμε αυτό. Βλέπουμε εδώ το 2016 είχαμε, ασχοληθήκαμε με τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων ειδικών συμβούλων, είχαμε την καθυστέρηση σε χημικές δοκιμασίες, Είχαμε την διεκπαιρέωση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των καταγγελιών παράβασης στο πλαίσιο του πιλωτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι καταγγελίες που λαμβάνουμε μας υποδεικνύουν πως ε, το πολιτικό πιλωτικό πρόγραμμα είναι πολύ αργό. Είναι κάτι επί του οποίου συνεχίζουμε να εργαζόμαστε. Έρευνε που κλείσαμε σε σχέση με το 2016 είναι η διαφανεία των τριμπερών διαλόγων, η πρόσβαση σε εκθέσει κλινικών μελετών σε σχέση με το Χουμίρα που είναι το προϊόν με τις ε, υψηλότερες πωλήσει στον κόσμο επειδή έχει αντιφλεγμονώδη δράση και πιστεύω πως χρησιμοποιήθηκε για τη δραματοειδή αρθρίτιδα νομίζω αλλά έχει επίσης δευτερεύουσες κρίσεις παραδείγματος χάρη σε σχέση με τη νόσο του κόν έτσι είναι πολύ πολύτιμο και σημαντικό για πολλούς ανθρώπους. Και αυτός, γι' αυτό και ασχοληθήκαμε με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων κλινικών μελετών. Επίσης με τις διαδικασίες της ΕΠΣΟ σε σχέση με ζητήματα αναθεώρησης. Και τέλος είχαμε τις στρατηγικές πρωτοβουλίες που ανοίξαμε το 2016 εδώ παραδείγματο χάρη ασχολούμαστε με ζητήματα όπω είναι έλλειψη διαφάνεια και το κατά πόσον άλλοι οργανισμοί εμπλέκονται σε σύγκρουση συμφερόντων ή κατά πόσον έχουν κώδικες δεοντολογίας. Η, επίσης ασχοληθήκαμε με τη διαφάνεια στο Eurogroup, το οποίο φυσικά και δεν είναι θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο έχουν ληφθεί πολλές πρωτοβουλίες για να γίνει πιο διαφανής η εργασία του και εμείς ενθαρρύνουμε την ε, πρωτοβουλία αυτή. Επίσης βρισκόμαστε σε διάλογο με την Ευρωπαϊκή Τραπεζα Επενδύσεων σε σχέση με το θέμα της διαφάνειας. Είχαμε τον πρόεδρο Χόιερ εδώ, με τον οποίο και συζητήσαμε σχετικά με το ζήτημα. Επίσης έχουμε την ε, διαδικασία αξιολόγησης και εποπτείας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και την προσβασιμότητά της, επίσης την προσβασιμότητα των ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανθρώπους με αναπηρίες. Εκεί μπορέσαμε και παρεμβήκαμε. Υπήρξε μια καταγγελία σε σχέση με αναπηρίες. Ήταν μια ενδιαφέρουσα καταγγελία επειδή δεν αφορούσε μόνο μια αναπηρία ακοής αλλά κάτι το οποίο πολλοί δεν αντιλαμβάνονται ότι άνθρωποι με προβλήματα ακοής χρειάζονται περισσότερο καιρό για να διαβάσουν ένα κείμενο. Οπότε σε εξετάσεις χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Είχαμε μία έρευνα σε σχέση με το κοινό καθεστώς υγειονομικής ασφάλισης για υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί ο ορισμός ήταν πολύ στενός Το επόμενο ήταν η προσβασιμότητα των ιστοσελίδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου, το Χουμίρα που ανέφερα πιο πριν, το συζήτησα σε αυτό το φόρουμ και σε άλλα, το ζήτημα του, της διάδρασης μεταξύ lobbying και δημόσιων υπηρεσιών. Συμβαίνει πολύ λόμπινγκ είναι κατανοητό και απαραίτητο και αναγκαίο. Κάποιες φορές όμως οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι σίγουροι για το πώς θα αντιμετωπίσουν το φαινόμενο, οπότε προβήκαμε σε μια δημόσια διαβούλευση και λάβαμε εξαιρετική ανάδραση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Συμβούλιο, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύσαμε έναν κατάλογο με πράγματα που θα πρέπει να κάνουν δημοσιοπαλοί και που δεν θα πρέπει να κάνουν, ντου και ντον, τη δύο στήλα στη διαφάνεια. Είναι ένας πρακτικός οδηγός, πιστεύουμε ότι θα είναι χρήσιμος για τους εκπροσώπους ώστε να γνωρίζουν των συμφερόντων, ώστε να γνωρίζουν κατά πόσον οι ίδιοι συμπεριφέρονται σωστά ή όχι. Πιστεύω πως με τον καιρό θα επικοδομήσουμε επί αυτού. Δεν θα εκπλαγείτε να το ακούσετε. Είναι κάτι ακόμα η διαφάνεια για τα δικαιώματα των πολιτών στη διαπραγματεύσεις περί Brexit. Ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησης. Αρχίσαμε αρκετά πρόημα με, την, με το θέμα αυτό. Επειδή πιστεύω πως μπορούμε να παίξουμε έναν πολύ χρήσιμο ρόλο όπως και το δίκτυο επειδή είμαστε όλοι άνθρωποι της... Εμείς όπως και η κοινωνία των πολιτών, οι συνθισμένοι πολίτες σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό θα επηρεαστούμε από αυτό που θα συμβεί τα επόμενα δύο χρόνια. Γι' αυτό και γράψαμε στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τους ρωτήσουμε για τα σχέδιά τους σε σχέση με την διαφάνεια και κατά πόσον θα υπάρξει διάλογος με προσώπους συμφερόντων και πολίτες. Ο πρόεδρος Γιούγκερ υποσχέθηκε τον Απρίλιο μια μοναδική και πρωτόγνωρη διαφάνεια. Τις τελευταίες εβδομάδες Είδαμε ήδη τη δημοσιοποίηση οδηγιών σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις. Φυσικά βρισκόμαστε ακόμα σε ένα πολύ πρόμοιο, πρώιμο εναρκτήριο στάδιο. Τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια θα συζητηθούν τα πραγματικά ευαίσθητα θέματα. Πιστεύω πως αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση που κάνουμε, καθώς αναμένουμε τις απαντήσεις του Συμβουλίου όπως και της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με αυτό που πρόκειται να γίνει. Παίρνουμε στη δεύτερη διαφάνεια. Εδώ έχουμε αυτή την ε, επιστολή του Γενικού Γραμματεία του Συμβουλίου. Στατική έρευνα, διαφάνεια στο Συμβούλιο και περίεργος το αποτέλεσμα όλη τη φασαρίας του Brexit είναι ότι οι πολίτε ενδιαφέρονται περισσότερο για το τι γίνεται στις Βρυξέλλες. Μεγαλύτερη επιθυμία να μάθουν. Κατά κάποιο τρόπο ε, τώρα προκάλεσε περισσότερο ενδιαφέρον. Κάποτε ο κόσμος ξέρει μόνο το, τους του, ήξερε ε, μόνο τους επιτρόπους του. Τώρα όμως αναγνωρίζει ας πούμε τον κύριο Γιούνκερ και επομένως θα πρέπει για το Συμβούλιο να έχει περισσότερη διαφάνεια γιατί θυμηθείτε τελευταία φορά λέγαμε ότι τίποτε δεν έχει υποβληθεί ως έτοιμο για το Συμβούλιο γιατί ο κόσμος τα βλέπει τα πράγματα από απόσταση θεωρεί ότι είναι πολύ αφηρημένος θεσμός στο Συμβούλιο επομένως θα είναι πολύ σημαντικά Άρα θα πρέπει να ανοίξει τις πόρτες του το Συμβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό. Και οι συνάδελφοι παρακολουθούν τι δημοσιεύεται, σε τι υπάρχει πρόσβαση, διαφορετικές μεθοδολογίες για τη διαφάνεια και για άλλα. Οπότε πρόκειται να διαμορφώσουμε κάποιες προτάσεις και να δούμε τι θα μας πούν τον Ιούνιο τώρα όσον αφορά τους τριμερείς διαλόγους έχουμε να κρεμεί απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το έγραφο με τις τέσσερις στήλες τον Ιούνιο δούμε τι απάντηση θα δοθεί επίσης ε, Πρόκειται να έχουμε επαφή με την κυρία Δίξτρον, όπως και πέρσι. Γιατί έχουμε αυτή την εκδήλωση και παλιότερα αυτά γινόντουσαν στις χώρες μέλη και είχαμε πολλά δίκτυα μεσολαβητών αλλά το τωρινό δίκτυο έχει ιδιαίτερη σημασία να είναι ευρωπαϊκό οπότε είναι σημαντικό να γίνει αυτή η εκδήλωση της Βρυξέλλες με τους αξιωματούχους Γι' αυτό και θεωρούμε ότι ε, είμαστε τυχεροί που θα έρθουν αυτοί οι ομιλητές που θα έρθουν Μέρι εκτός Βρυξελών. Θα συμμετάσχει και ο, ο ο δήμαρχος του Μέχελεν, που είχε το βραβείο του καλύτερου δήμαρχου στον κόσμο. Πολύ σημαντικό να ακούσουμε και εκείνο την άποψη. Θα είναι ο αντιπρόεδρος Τίμερμανς που θα κάνει την ε, καταληκτική ομιλία. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις. Thank you very much. And uh, some of those... Σας ευχαριστώ και κάποιοι, κάποια από τα θέματα αυτά που αναφέρετε ενδιαφέρουν πάρα πολύ τους συναδέλφους και είμαι βέβαιη γι' αυτό και εγώ θα ήθελα να συνεχίσουμε τη συζήτηση για κάποια από τα ζητήματα που αναφέρατε. Τώρα έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε και τους συναδέλφους. Η κυρία Μίτση είναι η συγγήτρια για την ετήσια έκθεση του 2016. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που έχασα το πρώτο τμήμα της παρουσίασής σας μου διαβιβάστηκε και ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ψήφιζα στι άλλε επιτροπέ. και είναι σημαντική η ψηφοφορία από ό,τι ξέρετε. Είμαι και βέβαια πολύ χαρούμενη που είμαστε και πάλι μαζί στην Επιτροπή Αναφορών. Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε. Κυρία μου που συνεργαζόμαστε. Ήμουν αρμόδια και για την έκθεση του 2015. Είναι χαρά και τιμή που συνεργαζόμαστε λοιπόν εκ νέου μαζί. Χαίρομαι που στην έκθεσή σας συνδέεται την εργασία των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και των ε, υπηρεσιών και της ε, εμπιστοσύνης που τρέφουν οι πολίτες προς την Ένωση και σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις που υπάρχουν ε, οι προκλήσεις που προκύπτουν από το μεταναστευτικό, από το Brexit, πρόκειται για προκλήσεις που αναφέρατε. Και αναφέρατε και από το που είναι ικανοποιημένοι οι πολίτες. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τους μηχανισμούς για την τόνωση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Αυτό θεωρώ ότι είναι και το μέλλον της ε, πολιτικής μας ζωής. Ο ρόλος του διαμεσολαβητή είναι πάρα πολύ σημαντικό και αναγνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι το έργο σας και πόσο καλά το επιτελείτε. Είσαστε πάντα προληπτικοί στη δράση σας. Αυτό είναι πραγματικά πολύ θετικό. Η διαφάνεια, ο ανοιχτός χαρακτήρας, η ταχύτητα ανταπόκρισης ε, μπορεί να βελτιωθεί. Τα έχετε όμως υπόψη σαν σας αυτά. Η έκθεση είναι στη διάθεσή μας ε, και δεν πρόκειται να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Έχω κάποιες ερωτήσεις να κάνω. Ο γενικότερος συντελεστής συμμόρφωση ε, σημειώνω σε ό,τι αφορά τι προτάσεις ε, της Ευρωπαία Διαμεσολαβήτριας έχει μειωθεί. Έχει μειωθεί αυτό ο συντελεστή. Από το 23% στο 19%. Γιατί, από πού προέρχεται αυτή η μείωση της συμμόρφωση, του παράγοντα συμμόρφωση. Είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε αυτό, γιατί δεν υπάρχει τώρα μεγάλη συμμορφώση. Θέλουμε φυσικά συμμορφώση 100%, αλλά αυτό είναι αδύνατο. Επίσης, 6,9% των περιπτώσεων κακοδιαχείρισης ε, το 2016 είναι, αυξήθηκαν σε 10,8%. πάλι μεγάλη διαφορά σε ό,τι αφορά την κακοδιαχείριση, αλλά θετική διαφορά αυτή τη φορά. Την αναγνωρίζουμε. Η διαφάνεια λοιπόν και πάλι. Το 2016 29,6 ήταν η διαφάνεια της 100. Αυτό αποτελεί κορυφαία ανησυχία όλων των πολιτών και νομίζω ότι εδώ έχουμε θέματα εμπιστοσύνης. Όταν υπάρχει διαφάνεια, θεωρώ ότι τονώνεται και η διαφάνεια. Και αυτό μας λείπει στα θεσμικά όργανα. Ένα τελευταίο ζήτημα. Το θέμα της χώρας προέλευσης. Ένα τμήμα των έρευνων αυτών ξεκινά στα κράτη-μέλη. Λίγες είναι όμω οι καταγγελίε εκείνες οι οποίες ξεκινούν από το γραφείο του διαμεσολαβητή. Γιατί? Αυτά είχα να σχολιάσω στην παρούσα φάση πριν ε, προετοιμάσω την έκθεσή μου και επίσης να σας επενέσω για τα πολύ καλά διαγράμματα που έχετε και τους παλούς, πολύ καλούς πίνακες. Είναι πάρα πολύ σαφείς. Κάτι άλλο, κάτι τελευταίο. 20% των καταγγελιών ολοκληρώθηκαν και έκλεισαν μετά από 18 μήνες, ενώ το, ο μέσος όρος είναι 12 έως 16 μήνες. Γιατί λοιπόν αυτό το 20% δεν κλείνει στο προβλεπόμενο αυτό διάστημα. Και τέλος να σας πω ότι προσβλέπω στην ε, κατάρτιση της έκθεσης και στη συνεργασία με τους ε, σκιώδεις. Ευχαριστώ, ο κύριος Βαλέτσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ σου το συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ εξ αρχής και εγώ ψήφιζα σε άλλη επιτροπή. Κάτι που θέλω να το πω γιατί με πνίγει. Είμαι μεγάλος φαν της κυρίας Ωραίλη Α, από την αρχή σας υποστήριζα. Προληπτικός, ε, δραστήριος ρόλος σας, σας θαυμάζω και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχετε τη θέση που έχετε. Να σας συγχαρώ επίσης για όσα έχετε κάνει για την καλή διαχείριση. Είναι πολύ καλή ιδέα και δίνει κίνητρα. Μου αρέσει επίσης το γεγονός ότι μετακινήσατε την ετήσια συνεδρίαση των αντιμεσολαβητών στις Βρυξέλλες πέρυσι και αυτό έχει νόημα. Για να έχουν την αίσθηση συμμετέχοντες το τι σημαίνει να λειτουργεί κανείς στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Και είμαι ευγνώμων που αναφερθήκατε στο θέμα του κράτους δικαίου στην Πολωνία πέρσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα αυτό και ελπίζουμε με τη βοήθειά σας να το επιλύσουμε. Προκειμένου η χώρα μου να μην είναι το παράδειγμα προς αποφύγη στην προκειμένη περίπτωση. Να σας συγχαρώ επίσης για το γεγονός ότι 70% των περιπτώσεων πέρσι ολοκληρώθηκαν μέσα σε ένα έτος. Πραγματικά εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ένα ερώτημα να κάνω όμως για το ποσοστό συμμορφωσή. 83% είναι το μέσος όρος. Αλλά υπάρχει μεγάλη απόκληση αναθεσμικό όργανο. Υπάρχει οποιαδήποτε τέτοιο οποιαδήποτε τέτοια εξήγηση για τις διαφορετικές αυτές ε, τα διαφορετικά αυτό αποτελέσματα ανά όργανο. Αυτά. Και σας ζητώ συγγνώμη αν δεν ακούσω την απάντησή σα, γιατί πρέπει σε 13 λεπτά να πάω σε ψηφοφορία τη Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου. Μα πολύ δύσκολε ημέρε, βαριέ, λέει η πρόεδρο. Ο κ. Μαριά. So... Θα μιλήσω ελληνικά. Ε, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την ε, Ombudswoman για την ε, σημαντική δουλειά που έχει κάνει. Άλλωστε και πέρυσι σαν ε, ραπορτέρ είχα την ευκαιρία να το εκφράσω αυτό και στο report. θεωρώ σημαντικά διάφορα ζητήματα που έχουν τεθεί. Η δραστηριότητα σε σχέση με την διαφάνεια που απαιτείται για το Eurogroup. Διότι το Eurogroup λαμβάνει τις πιο σημαντικές αποφάσεις αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει επιβάλει πολιτικές λιτότητας και έντονης ε, σκληρής δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει επηρεάσει τη ζωή των ίδιων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, το πρώτο βήμα που έγινε από την πλευρά της Κούμαν να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στις αποφάσεις του Eurogroup είναι ένα πρώτο βήμα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να επιμείνουμε κι άλλο ε, για να έχουμε ακόμη πιο σημαντικά αποτελέσματα. Να πω επίσης ότι ίσως πρέπει να θίξουμε και το θέμα των αποφάσεων του Eurogroup που εκδίδονται μόνο στην αγγλική γλώσσα την ώρα που οι αποφάσεις επηρεάζουν σημαντικά όλους τους λαούς, ιδίως στην Ελλάδα, και δεν υπάρχει μια επίσημη μετάφραση. Μόνο στα αγγλικά βγαίνουν οι αποφάσεις του Eurogroup. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Πέραν του ότι πρέπει να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στον κύριο Ντάισεμπρουμ για ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια στο Eurogroup. Δεύτερο, επιμένω στο θέμα που είχα θίξει και πέρυσι για τη σύγκρουση συμφερόντων που υπάρχει σε σχέση με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν μπορεί να είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ανεξάρτητη νομισματική αρχή και να εποπτεύει τις συστημικές τράπεζες και να είναι μέλος της Τρόικας και να είναι και δανειστής, ιδίως τώρα, με την ποσοτική χαλάρωση, το περίφημο QE. Επομένως, αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να το δούμε. Το δεύτερο είναι η ενημέρωση που κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για, το, την ποσοτική χαλάρωση. Έχω υποβάλει επανειλημμένα ερωτήσεις εάν συγκεκριμένες εταιρείες όπως είναι η Deutsche Bank ήταν ε, στις εταιρείες οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο αγοράς ομολόγων από πλευράς της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, το ίδιο συζητήθηκε και χθε, γιατί είχε έρθει ο κύριος Δράγκη και υπήρχαν συνάδελφοι από την Ισπανία, αν θυμάμαι καλά, που ρωτούσαν λεπτομέρειες για συγκεκριμένες ισπανικές εταιρείε που έχουν χρηματοδοτηθεί από την ποσοτική χαλάρωση. Δεν δίνει ενημέρωση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο θέμα αυτό και ούτε δίνει ακριβώς ε, λεπτομέρειες το τι ομόλογα έχουν αγοραστεί. Επομένως υπάρχει ένα θέμα διαφάνειας πολύ περισσότερο για την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία έχει δαπανίσει μέχρι στιγμής στην ποσοτική χαλάρωση για το 2015 και 2016 42,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δισεκατομμύρια ευρώ. Την ώρα που η Ελλάδα είναι εκτός ποσοτικής χαλάρωσης. Και ρώτησα να μάθω τι ομόλογα έχει αγοράσει. Και μου απήντησαν γενικώ και αορίστος. Αγόρασε ομόλογα του ESM, έχει αγοράσει η Τράπεζα της Ελλάδος ομόλογα του EFSF, αλλά δεν δίνουν λεπτομέρειες γιατί θέλω να δω πότε τα αγόρασε αυτά. Μήπως δηλαδή πρώτα αγόρασε τα ομόλογα του ESM και εν συνεχεία ο ESM δάνεισε την Ελλάδα. Δηλαδή μήπως η Ελλάδα έχει δανείσει τους δανειστές της και εν συνεχεία αυτοί δάνεισαν την Ελλάδα και επέβαλαν μνημόνια. Αυτό είναι κάτι που δεν μας το επιτρέπει, δεν μας δίνει τις απαντήσεις εν προκειμένου ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ε, η, Ευρω... Τράπεζα της Ελλάδος αγόρασε επίσης ομολόγα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πότε τα αγόρασε αυτά τι ποσό έδωσε. Διότι εν συνεχεία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έδωσε δάνειο στη Φραπόρτ η οποία άρπαξε τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να υπάρξει διαφάνεια. I'm going to finish, Madam Chair, ε, στο θέμα αυτό. Ε, το επόμενο ζήτημα, πολύ σύντομα βεβαίω, είναι ότι πρέπει να υπάρξει ακόμη σημαντική διαφάνεια στι διαπραγματεύσει για την TTIP και συγχαίρω την Ombudswoman για τι αποφάσει που πήρε πρέπει να δούμε τα διάφορα trade deals τα οποία γίνονται. Δεν αφορούν μόνο το Πακιστάν. Πρέπει να δούμε τι γίνεται στο Μπαγκλαντές, όπου αυτή τη στιγμή δεν τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, εργάζονται, τα παιδιά έχουν καεί, ε, οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια, ε, δεν υπάρχει καμία προστασία. Επομένως, για να κλείσω, θεωρώ σημαντική την έκθεση. Θα υποβάλω κι εγώ βεβαίως κάποιες τροπολογίες και να σας συγχαρώ άλλη μια φορά για την εργασία την οποία έχετε κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Άουκεν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή σας δουλειά και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχουμε εδώ την διαμεσολαβήτρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την έκθεσή σας. Δεν είναι πολύ βαριά στην ανάγνωση και ξέρω ότι καλύπτεται και περίπλοκες υποθέσεις. Να περάσω κατευθείαν στο ψητό. Καταρχάς, για το θέμα της διαφάνειας. Νομίζω ότι εδώ αντιμετωπίζουμε ένα κρυφό πρόβλημα και φυσικά το ξέρετε αυτό, ότι πρόκειται για μια διαρκή μάχη, ε, η οποία δύο βήματα μπροστά κάνει και δύο πίσω. Κάτι δίνουμε, κάτι χάνουμε. Το θέμα λοιπόν της διαφάνειας και στη δική μου τη χώρα ε, είναι ένα θέμα. Έχουμε το θέμα όμως της ε, έλλειψη διαφάνεια για την ΕΦΣΑ, για την έκθεση για την κλεφωσάτη. και έχουμε μείνει πίσω. Δεν έχουμε ευκαιρία να ρωτήσουμε τους υπηρεγνώμονες μας τι γίνεται με την αξιοποίηση αυτή, με την εξολογήση αυτή. Αυτό θεωρώ ότι υπονομεύει την δουλειά μας. Ξέρω ότι κάνετε ό,τι μπορείτε, αλλά νομίζω ότι καλά θα κάνουμε να τονίσουμε ακόμα πιο πολύ ότι τα σώματα λήψη αποφάσεων είναι απόλυτα υποχρεωμένα να έχουν καλή διαχείριση και διαφάνεια. Ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και γιατί βλέπω ξανά και ξανά ότι τα σώματα αυτά δεν μιλώ για πολιτικές υπηρεσίες αλλά για διοικητικές υπηρεσίες με μια απλή δήλωση ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, τη βγάζουν καθαρή. Και μετά ακούμε από, το, από τον Δανό διαμεσολαβητή ότι σε καμία περίπτωση δεν μας πρέπει να μας ικανοποιεί αυτή η δήλωση έλλειψη σύγκρουση συμφερόντων, γιατί πολύ απλά δεν δηλώνονται τέτοια ζητήματα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια διαρκή μάχη. Γιατί το έθεσα και στον Τίμερμαν, αλλά μπερδεύτηκε στην απάντησή του. μπλέχθηκε με το θέμα του revolving doors, αυτής της ε, διαδοχικής ε, ανάληψης καθηκόντων ε, από πολιτικά πρόσωπα σε επιχειρηματικές επιχειρήσεις. Και το θέμα της διαφάνειας. Το Συμβούλιο. Αυτή η έλλειψη διαφάνειας που επικρατεί στο Συμβούλιο είναι κάτι που βαραίνει πάρα πολύ τα εθνικά κοινοβούλια. Στο Δανικό Κοινοβούλιο, για παράδειγμα. Πρόκειται για μία από τι πιο παλές ε, Ευρωπαϊκές Επιτροπές, Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και δεν έχουν πληροφορίες σωστέ από το Κοινοβουλίο για το τι γίνεται στο Συμβούλιο. Δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν. Πώς να ξέρει πώς να συμπεριφερθεί η ιδανική κυβέρνηση, το ιδανικό κοινοβούλιο, ήταν ε, η ιδανική κυβέρνηση δεν έχει καν τι θέσει που χρειάζεται. Αυτή η έλλειψη διαφάνεια στο Συμβούλιο μας δυσκολεύει πάρα πολύ και στους τριμερείς διαλόγους. Γιατί αν η μία πλευρά είναι διαφανής και η άλλη είναι τελείως διαφανής, άμα τι θα γίνει. Δεν λύνονται τα προβλήματα. Χρειάζεται πολύ παραπάνω διαφάνεια, όχι μόνο για το έργο του Κοινοβουλίου, αλλά και για τους πολίτες και για τη δυνατότητα να παρακολουθούν το τι συμβαίνει σε δημοκρατικά θεσμικά όργανα. Υπάρχει ένα δημοκρατικό σύστημα. Αλλά φαίνεται ότι οι πολιτικοί δεν έχουν πραγματικά κινητοποιηθεί, δεν έχουν αξιοποιήσει αυτό το δημοκρατικό σύστημα. Και εδώ η έλλειψη διαφάνειας είναι που κάνει τη διαφορά. Δεν ξέρω κατά πόσον σα απασχολεί στην έκθεση αυτή, τουλάχιστον με το βλέπω να σας απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα της έλλειψης διαφάνειας στο Συμβούλιο. Δεν είναι θέμα μόνο πολιτικών λόμπι. Το θέμα είναι και τι συμβαίνει τελικά στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λεκή πρόεδρο. Κύριε Μπεσέρα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Από πλευρά του κύριου Νάρτ είναι για τους ελεύθερους συνεισηγητής. Ευχαριστούμε κύριε Ράιλε για την εκθεσή σας. Ευχαριστούμε για το έργο σας. Η Άλντε θα βοηθήσει με κάθε μέσον το έργο σας. Τρέχουμε μεγάλο σεβασμό για τον ρόλο τον οποίο διαδραματίζεται και για τη βοήθεια προς την Επιτροπή των Αναφορών. Εγώ είμαι συντονίστρια για την Άλντε στην Επιτροπή μας. Θα σας ε, βοηθήσω, αναγνωρίζω τους προσπαθειές σας, ε, νομίζω ότι βοηθάτε πάρα πολύ και αυτοί που σας θαυμάζουν, οι φαν, συνέχεια αυξάνουν την περασμένη εβδομάδα, είδατε τι έγινε ε, για την εκδήλωση που αφορούσε το τι θα γίνει το δικαιώματα των Ευρωπαίων στη Βρετανία. Είχαμε, έχουμε 100.000 Ισπανούς στην ε, ε, Ισπανία. Επίσης είπαμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το δίκτυο των ε, διαμεσολαβητών. Είπαμε ότι θα πρέπει από κοινού να προχωρήσουμε στην διεκπαιρέωση των αναφορών για το Brexit. Θα πρέπει να προσέξουμε το ότι θα εποπτεύουμε κάθε προσπάθεια τον υπάρχει περισσότερη διαφάνεια και για τα έγγραφα, την προσβασιμότητα στα έγγραφα ε, και τη δημοσιότητα που δίνεται σε διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις. Ανησυχούμε σε σχέση με το ότι δεν υπάρχει προσβασιμότητα σε κάποια έγγραφα που αφορούν τις παραβιάσεις της ελεύθερης κυκλοφορίας από πλευράς Ηνωμένου Βασιλείου και τις σχετικές αγωγές που έχουν γίνει. Έχουμε πάνω από 400 Ευρωπαίους που μας έχουν γράψει σχετικά με αυτές τις παραδιάσεις του κοινωτικού δικαίου. Θα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή των καλών πρακτικών, ε, θα πρέπει να ε, πέσει άπλο το φως αυτά τα οποία γίνονται σωστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης και, για τα βραδεία που είπατε και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Θεσπίσατε ένα προηγούμενο και εμείς λέμε να συνεχιστεί αυτή η πορεία. Να μαθαίνει το πόσο απαραίτητη η Ευρωπαϊκή Ένωση ο κόσμος. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Είναι το λόγο στην κυρία Εύη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμότατα κύριε Διαμεσολαβήτρια για όσα κάνετε πραγματικά έτσι καταφέρνετε να γίνεται κάτι για αυτά τα σοβαρά προβλήματα που έχει η Ευρώπη. Είπαμε επίση και για κάποια κενά που υπάρχουν στη δουλειά μας, ε, για πάρα πολλούς τομείς, όπως τα περιγράψατε σήμερα και τα επισήμεναν και συνάδελφοι, οπότε να μην τα επαναλάβω τα όσα ακούσαμε. Θα πρέπει να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα, να αποκτήσουμε έτσι ξανά αξιοπιστία. Πάντως, κάτι άλλο θα πρέπει να προσέξουμε, είναι κάτι το οποίο αποτελεί περιεχόμενο απαντήσεων από τα θεσμικά όργανα. Ιδίω όσον αφορά όταν, τι γίνεται όταν πιέζουμε τα θεσμικά όργανα για διαφάνεια, για τους ειδικού συμβούλους, για οικονομικά συμφέροντα, για τους τριμερείς διαλόγους, για όλα αυτά. Όπως και οι συνάδελφοι που μίλησαν πριν, θέλω να πω ότι επήγει το ζήτημα να μπορέσουμε να αναλάβουμε δράση και να μπορέσουμε να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα, να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων. Τώρα να σας αναδείξω κάτι το οποίο συμβαίνει από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόκειται για κάποια υπόθεση που αφορά πολλές αναφορές που έχουμε λάβει στην Επιτροπή μας. Έχουμε τέσσερις αναφορές ανοιχτές και αφορούν κάποιο είδου καταχρηστική χρήση συμβάσεων εργασίας στην Ιταλία. Και έτσι η οδηγία 99 του 70 παραβιάζεται. Έχουμε πολλές τέτοιες καταγγελίες, πολλές έρευνες και έχουμε και πολλές αγωγές επί παραβάση κατά της Ιταλίας. Και έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις στον τομέα της δημόσιας παιδείας. Η Κομισιόν τι λέει. Έχει πει πολλές φορές ότι δεν είναι παραδεκτές οι αναφορές, ε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε άλλους ε, τομείς κρατικής δραστηριότητας και όχι μόνο στη δημόσια παιδεία και λέει ότι θα πρέπει να εξετάζουμε τι ισχύει στο σύνολο του δημοσίου. Έχουμε το ίδιο Pilot του 2013. Έχουμε μόνο ένα σωρό αγωγές κατά της Ιταλίας και είπαμε ότι θα πρέπει να εξεταστεί πώς συνολικά διεκπεριώνει αυτά τα προβλήματα η Επιτροπή. Μα αργεί πάρα πολύ, καθυστερεί. Έχουμε διαδικασία EU Pilot και είπαμε ότι χρειάζεται πολλές φορές δεύτερη διαδικασία επί Και το Δεκέμβριο του 2015 τελικά αποφάσισε η Επιτροπή τη μία από αυτές να την αρχιοθετήσει. Και η Ιταλία ανέλαβε να θεσπίσει ένα νέο νομοθέτημα για το προβληματικό σημείο. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει καλύτερος έλεγχος από την Επιτροπή. Θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους να δούμε κατά πόσον αποδίδει αυτό το νέο νομοθέτημα γιατί θίγονται πάρα πολλοί εργαζόμενοι στη δημόσια παιδεία. Δεν θα πρέπει αυτού του είδους συμβάσεις εργασίας να χρησιμοποιούνται καταχρηστικά. Άρα, έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και από την Κομισιόν και από τις Ιταλικές Αρχές. Χρειάζεται επομένω πιο δυναμική παρέμβαση. Έχουμε εδώ μια περίπτωση κακοδιοίκησης. Πρέπει να υπάρξει περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη στοιχεία γιατί χιλιάδες ανθρώπων φύγονται. Η κυρία Εσταράς. Συγχαρητήρια προς τη Διαμεσολαβήτρια για το έργο της. Συμφωνώ με όσο είπαν οι συνάδελφοι και εγώ θέλω να σας πω κάτι για αυτό το οποίο συζητούμε εδώ στο Κοινοβούλιο όσον αφορά την προσβασιμότητα. Δεν σας έχει απασχολήσει βέβαια ακόμα, αλλά με την ευκαιρία θέλω να σας πω ότι αυτή, αυτό το νομοθέτημα για την προσβασιμότητα πλευράς των αναπήρων ε, πασχόλει πάρα πολλούς φορείς αυτών των προσώπων και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς και να δούμε τι θα γίνει με το νομοθετήμα. Όπως ίσως θυμάστε, η Επίτροπος Ρέντινγκ έχει κάνει τη σχετική εξαγγελία. Ε, εμάς μας ενδιαφέρει πολύ, έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις και επίση το αντίστοιχο όργανο του ΟΗΕ ε, ασχολείται με αυτό το θέμα. Τελικά η Επίτροπος ε, Τάισεν έκανε κάποια πρόταση που εγκρίθηκε, αλλά τελικά ε, συνέχισε να ασχολείται η ΙΜΚΟ. Η ΙΜΚΟ είναι η Επιτροπή που ασχολείται με τις επιχείρησεις. Δεν θα έπρεπε να αναφέρει αυτό το, το, θέμα το οποίο απασχολεί και τόσο πολύ τους αναπήρους. Ε, εμείς επομένως έχουμε ένα σωρό επαφές με τους ενδιαφερόμενους όπως είναι σήμερα το σχέδιο ε, αυτού του νομοθετήματος δεν λέει τίποτα. Γι' αυτό και ε, έχουμε λάβει πάρα πολλές αναφορές, τις έχουμε διαβιβάσει, ε, λέτε για εξαίρεση των μικροεπιχειρήσεων, λέμε για προσβασιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, για τα, για τα κτίρια σε πολλά κράτη-μέλη παρά το δίκαιο ε, παρά τους νόμους που υπάρχουν ούτε εκεί υπάρχει προσβασιμότητα ε, αυτό αφορά ακόμα και τα ATM και, και αυτά θα έπρεπε να ε, είναι προσβάσιμα τι γίνεται επίσης με τηλεοπτικές εκπομπές τι γίνεται αν μπορούν να τα ακούσουν να έχουν προβλήματα ακοής ε, που τι μπορεί να γίνει, τι εκπομπές που υπάρχουν. Δηλαδή, αυτή η οδηγία τελικά δεν ωφελεί τους αναπήρους, ωφελεί τη βιομηχανία. Η Επίτροπος κυρία Τίσεν ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το θέμα. Μιλάμε για μια επταετία που έχει ε, χρονίσει αυτό το μέτρο. Οι φορεί των απείρων ε, είναι πάρα πολύ οργισμένοι. Θα πρέπει εμάς να μας πείτε τι μπορεί να κάνετε. Κυρία Ροζιέρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την διαμεσολαβετρία ε, για την παρουσίαση και για την έκθεση της να τονίσω τον κέριο ρόλο που παίζει και κυρίως ε, σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και τον δημοκρατικό χαρακτήρα των ε, οργάνων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν για το ρόλο που παίξετε. Κατά τον ίδιο τρόπο σε ό,τι αφορά την έρευνα για τον κώδικα δεοντολογία, σε ό,τι αφορά τη δήλωση ελεψής σύγκρουσης συμφερόντων, πρόκειται για πρωτοβουλίε εξαιρετικά α, πραγματικά. Σας ενθαρρύνουμε λοιπόν να συνεχίσετε στον ίδιο δρόμο. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα συγκεκριμένο θέμα ωστόσο το οποίο μας απασχολεί εδώ στο Κοινοβούλιο και κυρίως στην Επιτροπή Δυναμικών Υποθέσεων ό,τι αφορά ε, σε ό,τι αφορά το θέμα του συναγερμού σε ό,τι αφορά τον ρόλο του συναγερμού, σε ό,τι αφορά δραστηριότητε ε, που έχουν σημειωθεί στα πλαίσια του Κοινοβουλίου για φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή. Ολοκληρώσονται το 2015 μια σχετική έρευνα για το ότι δύο μόνο από τα 11 όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν ε, ακολουθήσει τις συστάσεις σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά για την ε, ειδοποίηση. Έχετε ωστόσο σημειώσει καμία άλλη πρόοδο σε ό,τι αφορά αυτή την ειδοποίηση. Γιατί η έκθεση του 2016 δεν συνέχισε, δεν παρακολούθησε το θέμα αυτό, θεωρείτε ότι ολοκληρώθηκε με τις συστάσεις του 2015. Σε κάθε περίπτωση το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί τα θέματα αυτά και θα ήθελε να παρακολουθήσει τα θέματα αυτά και σας ευχαριστώ εκ του προτέρων για την απάντησή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ντάρλινγκ, η οποία και ολοκληρώνει τον κατάλογο των ομιλητών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα συγχαρώ και εγώ την διαμεσολαβητρία για τη δουλειά της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία και με το Κοινοβούλιο. Δύο μόνο στοιχεία από δική μου πλευρά τα τελευταία χρόνια. Έχετε κάνει πολλά για την εμπορική πολιτική λόγω και των σκανδάλων που ξέσπασαν για τις διαπραγματεύσεις, για το TTIP, για την έλλειψη διαφάνειας στις εμπορικές συμφωνίες. Φαίνεται ότι τα φώτα των προβολέων έχουν πλέον μετακινηθεί, μια και έχει παγώσει πλέον το TTIP, ενδεχομένω να αναθερμανθεί με τον Τραμπ. Ποιο ξέρει κιόλα. Αλλά στην παρούσα φάση το θέμα έχει βγει από το ραντάρ. Εκ παραλλήλου γίνονται και μεγάλε εμπορικέ διαπραγματεύσει, οι οποίε γίνονται λίγο εκτό ε, τη ζώνη ε, του ραντάρ. Ακούμε πολλές ανησυχίες για την συμφωνία με την Ιαπωνία έχουν εκφραστεί λοιπόν πολλές ανασυχίες, αλλά δεν έχει παρακολουθηθεί τόσο πολύ το θέμα αυτό από τη δημοσιότητα. Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να σα παρακαλέσω το εξή. Όχι επειδή δεν πρόκειται για το TTIP και δεν είναι σεξ το θέμα, να σταματήσουμε να παρακολουθούμε τα θέματα των εμπορικών συμφωνιών. Γιατί το θέμα του TTIP ε, το προωθήσατε αρκετά και γι' αυτό το παρακολουθήσαμε. Για το Brexit, κατά δεύτερον, να σας ε, απευθύνω μια έκκληση σε ό,τι αφορά τους ε, πολίτες της Βρετανίας που θα χάσουν την ηθαγένειά τους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εμείς από βρετανικής πλευράς δεν έχουμε από πλευράς της κυβέρνησης μας διαφάνεια για το τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις και αυτό προφανώς προκαλεί όλο και μεγαλύτερη ανησυχία και εκνευρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και το θέμα λοιπόν του Brexit και το θέμα της διαφάνειας για τις διαπραγματεύσεις του Brexit να έχετε υπόψη και το σκέλος ε, των Βρετανών πολιτών που θέλουν διαφάνεια για τις διαπραγματεύσεις. Πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, όντως, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Οράιλε για να απαντήσει στις ερωτήσεις που ετέθησαν. Και παρακαλώ, αν δεν θέλετε να επισέλθετε σε λεπτομέρειες, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, υπάρχει η δυνατότητα να απαντήσετε γραπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε και φυσικά το ίδιο θα πω και σε οποιονδήποτε θέλει να επισέλθει σε λεπτομέρειε για οποιοδήποτε θέμα το οποίο ακούσαμε σήμερα, να γίνει αυτογραπτά γραπτά δηλαδή. Σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση, κυρία Πρόεδρε. Πέρσι είχαμε 19%. Ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι βέβαια, αλλά ξέραμε ότι θα ήταν προβληματικό αυτό, γιατί το 90%, το 90% ε, δεν θα μπορέσαμε να το ξαναπετύχουμε. Το 83% ήταν το, καλύτερο αποτέλεσμα, το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της υπηρεσίας. Για τη διαφάνεια επίσης και ακούσαμε και το θέμα της διαφάνειας του λόμπι για τον καπνό, το οποίο και απορρίφθηκε, ήταν πάρα πολύ κρίσιμο τότε σε σχέση με τις στάσεις και τις καταγγελίες γενικά. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που έχω που κάνω τις στρατηγικέ έρευνες είναι ότι αυτό βοηθά ακόμα και εκείνους που δεν έχουν άμεσες σχέσεις με τα θεσμικά όργανα και δεν γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται. Κύριε Βαλέσα, για την ε, καλή διαχείριση και πάλι να σας πω ότι αυτό ήταν ρηψοκίνδυνο γιατί ρηψοκινδυνεύουμε αυτό το βραβείο που δίδεται σε μια υπηρεσία, τελικά η υπηρεσία αυτή έκανε να κάνει κάτι τραγικό στη συνέχεια. Δεν έχει συμβεί αυτό. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή εκδήλωση αυτή και ήταν τρόπο όχι μόνο να προαγάγουμε τι βέλτιστε πρακτικέ, αλλά να προβάλλουμε και εξαιρετικό έργο κάποιων υπηρεσιών ή συνεργασία υπηρεσιών σε ό,τι αφορά τώρα το Eurogroup και τη διαφάνεια του Eurogroup. Έχω δουλέψει από αυτό. Πρόκειται για μια εργασία η οποία βρίσκεται εν εξελίξη και το παρακολουθώ το θέμα αυτό συνεχώς ε, και το θέμα των ομολόγων. Ξέρω ότι και το Κοινοβούλιο κάνει πολλή δουλειά επ' αυτού και πολύ υποπτεύομαι ότι όλη αυτή η δουλειά του Eurogroup για το μέλλον ε, και τη διαφάνεια των εργασιών της θα ε, επικεντρωθεί ιδιαίτερως όταν τελειώσουν και οι γερμανικές εκλογές, γιατί ήδη γίνεται μεγάλη πολιτική συζήτηση για το θέμα αυτό και σίγουρα θα το εξετάσουμε ε, Ιδιαίτερο όχι το πολιτικό σκέλο αλλά το διοικητικό σκέλο. Το έχω υπόψη μου και για την κυρία Άουκεν σε ό,τι αφορά την έκθεση για την γλυφοσάτη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο οι πολίτε να τα ξέρουν αυτά. Να ξέρουν ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας λέει ότι εντάξει, η ΕΦΣΑ να λέει το αντίθετο. Η ΠΟΗ να αποφαίνεται ότι ενδεχομένω να υπάρχει κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και πάλι η ΕΦΣΑ να αρνείται. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να σας πω, άλλο σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και πάλι. Προφανώς τα σχόλιά μου είναι προφανή. Στη Δανία δεν είσαστε βέβαιοι τι γίνεται με τους Δανούς πολιτικούς. Και αυτός νομίζω ότι αποτελεί μια κατάσταση που ισχύει σε αρκετά κράτη-μέλη. Επίσης, και αυτό μου το επεσήμαναν και Άγγλοι βουλευτές που μας είπαν ότι δεν ξέρουν τι πράττουν οι, οι υπουργοί τους. Η λογοδοσία όμως ε, προς όλους τους μεμονωμένους λαούς ε, αποτελεί ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το κοιτάξουμε σε το κρατών μελών. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα τις έρευνές μας αυτές για τη διαφάνεια του Συμβουλίου. Αυτό που κάνουμε από τις ομάδες εργασίας ε, μάλλον είναι ένα μεγάλο κομμάτι δουλειάς που αποτυπώνει, θεωρούμε, καλά το πολιτικό σκέλος της δουλειάς, το οποίο το έχουμε υπόψη μας ε, τώρα, σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις επί παραβάση και τα πολιτικά προγράμματα τα οποία εξετάζουμε. Λαμβάνουμε πολλές καταγγελίες και πάλι το έργο αυτό για το πολιτικό σύστημα θα έπρεπε να διευκρινίζει ζητήματα για την διαδικασία σε επιπαραβάση. κυρία Ήδη σε ό,τι αφορά τι περιπτώσει και τι καταγγελίε που αναφέρατε, τι γνωρίζω, τι έχω υπόψη μου. Νομίζω ότι πλέον υπάρχει απόφαση δικαστική κομισιόν κατά τη ναι. σχετικής ε, κυβέρνηση. Εγώ δεσμεύομαι να μην συμμετέσχω, να μην παρέμβω σε περίπτωση δικαστική απόφαση Όταν δημοσιευτεί η δικαστική απόφαση θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να με τηρήσει ενήμερη σχετικά με το τι προτίθεται να κάνει. Προ το παρόν έχει παγώσει λοιπόν το θέμα αυτό μέχρι ότου να αποφανθεί το δικαστήριο. Αλλά σίγουρα το παρακολουθώ το θέμα. Προφανώ, ε, σε ό,τι αφορά το θέμα τη αναπηρία. Η πραγματική απάντηση είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση. Εγώ μπορώ να κάνω τη δική μου δουλειά, αν θέλετε, να συλλέξω τι καταγγελίε κτλ. όπου υπάρχει ζήτημα για την αναπηρία. Αλλά η πολιτική οι πρωταθλητέ από τον τομέα τη πολιτική, όπω εσεί θα είναι αυτοί που θα προωθήσουν το θέμα αυτό και τι καταγγελίε αυτέ. Και η κυρία Ρουδιέ έθεσε το θέμα των ε, πληροφοριοδοτών, των whistleblowers. Αυτό το θέμα είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και το 2016 ενδεχομένως να μην είχαμε ακόμα τα κατάλληλα στοιχεία στη διάθεσή μας για να αντιδράσουμε. Θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε για να δούμε πώς εφαρμόζονται στην πράξη αυτοί οι κανόνες για την προστασία του. Για την κυρία Ντάρλινγκ, Κέρτιν Ντάρλινγκ. Ναι, πριν από τρει εβδομάδε ήμουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο, που σφίζει από κόσμο δεν υποφέρει ακόμα από τον Brexit και συναντήθηκα με τη Σχετική Επιτροπή Ενημέρωση για να συζητήσω ακριβώ το θέμα αυτό. Την πρωτοβουλία. Και θα ήθελα να μιλήσω λοιπόν με την αρμόδια αν υπήρχε πρόβλημα σε ό,τι αφορά α, την παροχή πληροφοριών από την ε, Βρετανική κυβέρνηση, θα μπορούσαν να ζητήσουν τα αρχεία αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πολλά από τα αρχεία αυτά θα τηρούνται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολίτε του Ηνωμένου Βασιλείου θα έχουν ίδιο δικαίωμα πρόσβαση στα έγγραφα αυτά, όπω και οι υπόλοιποι πολίτε. Εγώ από πλευρά ε, του δικού μου τη δική μου υπηρεσία θα πρέπει να σα πω ότι θα συνεχίσουμε να απασχολούμε του εξαιρετικού Βρετανού συναδέλφου ε. αν ναι, υπάρχει θέμα έλλειψης διαφάνειας από πλευράς της Βρετανικής κυβέρνησης, πάντα μπορούν οι πολίτες του, του Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. Εξαιρετική, εξαιρετική απάντησή σας και η παρουσίασή σας, λέει η Πρόεδρο. συγχαρητήρια σας. Γιατί απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, όπως πάντα άλλωστε, οι ανακοινώσει που έχω λοιπόν για σήμερα. Στις 11 Ιουλίου έχουμε την εξέταση της έκθεσης. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 11 Ιουλίου. Ωραία, 3 το μεσημέρι. Α, όχι. 18 Ιουλίου, λάθος, Πέτρος. 3 το απόγευμα, προθεσμία. Θα ψηφίσουμε 10 Οκτωβρίου του 2017. Ναι. Και θα πάμε στην Ολομέλεια το Νοέμβριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και καλό κουράγιο για να ανταποκριθείτε στις ανάγκες των πολιτών της Ευρωπαϊκή Ένωση, των 28 ακόμα κρατών μελών. Okay, and uh, the petitioners are here. I am εντάξει, οι αναφέροντες είναι εδώ. Λυπούμε που σας έκανα να περιμένετε λίγο, επειδή έχουμε ένα σημείο ακόμα στην ημερήσια διάταξη που είναι η διερευνητική επίσκεψη στη Μαυρίτη. Πρέπει να το εξετάσουμε πρώτα. Ο επικεφαλής της αποστολής βρίσκεται εδώ. Θα μας ενημερώσει σύντομα για την επίσκεψη. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ήμασταν μια αποστολή πέντε ανθρώπων στη Μαδρίτη την περασμένη Δευτέρα και Τρίτη. Συνοδευτήκαμε από τρία αυτεπάγγελτα μέλη από την Ισπανία το οποίο μας έκαναν μια ευμεγεθή αποστολή ήταν μια, πολύ, μια επίσκεψη με πολύ πυκνό πρόγραμμα όχι μόνο λόγω του θέματος αλλά επίσης λόγω του χρονοδιαγράμματος, του αριθμού των συναντήσεων που είχαμε όσο ήμασταν εκεί. Οπότε ασχοληθήκαμε με αναφορές που αποτελούν σκάνδαλο ότι χιλιάδες να εστάλησαν από νοσοκομιακό προσωπικό σε πολλές περιπτώσεις από εκκλησιαστικά νοσοκομεία κατά τη δικτατορία στην Ισπανία τα οποία διατέθηκαν για υιοθεσία από τη δεκαετία του 40 έως τη δεκαετία του 90. Είχαμε συναντήσεις με τον Ισπανό Υπουργό Δικαιοσύνης, με τον εκεί διαμεσολαβητή και τον αναπληρωτή διαμεσολαβητή, με την Ισπανική Καθολική Εκκλησία, με ενδιαφερόμενους δημοσιογράφους, αλλά και με τα θύματα τα ίδια συμπεριλαμβανομένου ενός πολίτη του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος προσδίδει μια πιο ευρωπαϊκή διάσταση στις περιπτώσεις αυτές, καθώς είναι μη Ισπανός πολίτης. Οπότε μπορώ να παρουσιάσω εδώ κάποιες από τις εντυπώσεις μας από την επισκέψη της περασμένης εβδομάδας είδαμε αντιφατικά στοιχεία, προφανώς αντιφατικά στοιχεία από αυτούς που εκπροσωπούσαν δημόσιες αρχές σε σύγκριση με αυτούς εκ των έξω, θύματα και αυτούς που εκπροσωπούσαν τα θύματα ή αυτούς που μιλούσαν ως ακτιβιστές, δημοσιογράφοι, δικηγόροι. Για να καταλάβετε το μέγεθος του σκανδάλου, οι αριθμοί διέφεραν εντελώς που μας έδιναν επίσης το κατά πόσο μιλούσαμε για μεμονωμένα περιστατικά ή κατά πόσον εννοούσαμε ένα οργανωμένο κύκλωμα εμπορίας νεογνών. Ήταν ξεκάθαρο πως οι δημόσιες και εκκλησιαστικές αρχές δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τα θύματα. Τα θύματα και οι αναφέροντες πρέπει να περάσουν να πληρώσουν κάποιες προϋποθέσεις για να θεωρηθούν θύματα. Πρέπει να αποδείξουν οι ίδιοι τις περιπτώσεις τους και πολλές φορές επί δεκαετίες αναγκάστηκαν να διερευνήσουν το παρελθόν τους με λίγη καθόλου ψυχολογική υποστήριξη. Αυτά μέχρι που ξέσπασε το σκάνδαλο το 2009-2010. Τότε είχαμε εξελίξεις. Εκεί είχαμε ένα γραφείο υποστήριξης θυμάτων κατά την πρόσβασή του στα αρχαιακά έγγραφα. Με όσους μιλήσαμε αναγνώρισαν πως έγιναν πολλά για να βελτιωθεί η κατάσταση των θυμάτων. Το τελευταίο συμπέρασμα που έχω είναι αρκετά πολιτικό, αλλά είναι σημαντικό να υποθεί πως κατά βάση αυτό που ήταν ξεκάθαρο είναι πως το σκάνδαλο αυτό είναι το χειρότερο μέρο των πληγών του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου που δεν έχουν επουλωθεί ακόμα. Αυτό ήταν σαφές, πολύ σαφές κατά την επίσκεψή μας. Είχαμε κάποια βήματα προς τα μπροστά, τα οποία επικροτήσαμε και είδαμε την περασμένη εβδομάδα. Κανείς δεν είπε ότι δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα. Αυτό είναι μια βελτίωση. Η συνάντηση με την Εκκλησία ήταν πολύ θετική. Η Εκκλησία συμφώνησε να ανοίξει τα αρχεία της. Τώρα πρέπει να διασφαλίσουμε πως στις, στα λόγια θα ακολουθήσουν πράξεις. Και μία πρόταση ήταν να συνδέσει η Εκκλησία τα ιδιωτικά αρχεία της με τα δημόσια αρχεία του Γραφείου Υποστήριξης Θυμάτων. Και η τρίτη, το τρίτο θετικό βήμα ήταν οι ειδήσει πως εθνικοί βουλευτές ζήτησαν τη σύσταση μιας κοινοβουλευτικής διερευνητικής επιτροπής για το θέμα επειδή Υπάρχει μεν η προσέγγιση από περίπτωση σε περίπτωση, αλλά υπάρχουν τόσο πολλέ ομοιότητες που μπορεί να υπάρξει και μια ομαδική προσέγγιση. Τώρα ε, καταρτίζουμε την έκθεση, η οποία μπορεί να διαφέρει από τις δικές μου προσωπικές εντυπώσεις, αλλά πιστεύω πως συλλογικά θα μπορούσαμε να παίξουμε τον ρόλο μας, αντιμετωπίζοντας τις ανησυχίες των αναφερόντων και να χρησιμοποιήσουμε την επισκεψή μας για να ασχοληθούμε επικοδομητικά με το θέμα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι μια ευκαιρία να ακούσουμε, δεν είναι η στιγμή για μια συζήτηση, ακούμε μόνο, ακολουθούμε τους κανόνες, ακολουθούμε μόνο τις εντυπώσεις από μια διερευνητική επίσκεψη, συζήτηση θα γίνει μόνο αφότου υποβληθεί κείμενο. Η συζήτηση έγινε την περασμένη εβδομάδα, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα συζητήσουμε επί αυτής τώρα. Επίσης έχουμε κάποιο που πρέπει να αποχωρήσει από το χώρο σε λίγα λεπτά. Οπότε τον Ιούλιο ή τον Σεπτέμβριο θα εξετάσουμε το έγγραφο κείμενο και τις συστάσεις. Αυτό δεν ήταν παρά μια παρουσίαση ενώπιον όλης της Επιτροπής, γι' αυτό και Γιού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδα ήδη σήματα από δύο συναδέλφους, γνωρίζω πως αν αρχίσω τη συζήτηση τώρα θα χαθούμε το οποίο σημαίνει πως δεν θα γίνει συζήτηση τώρα, θα προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι οι αναφέροντες. Συγγνώμη για αυτό, αλλά πρέπει να είμαι δίκαιη. Ευχαριστώ πολύ Τζουτ που μας έδωσες μία εκ των για το ταξίδι αυτό και θα εξετάσουμε το κείμενο αυτό όταν το παρουσιάσεις. Θα ήθελα να μισώ εδώ το λόγο. Όχι, όχι, όχι, δεν γίνεται γιατί δεν θα γίνει συζήτηση. Ναι, αλλά δεν συμφωνώ με αυτό που ανεφέρθη. Ταυτόχρονα μιλάει και ο κύριος Μαριάς, θα δεν ακούγεται. Ήμουνα και εγώ στην αποστολή. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Ε, κάτι προσωπικό είπε η πρόεδρος, θα πρέπει αυτό να αποκατασταθεί. Ήταν προσωπική πρόεδρο. Η πρόεδρος λέει ότι αν σας δώσω το πρέπει να το δώσω σε όλους. Όχι, Πρόεδρε, πρέπει να μου το λόγο, γιατί έκανε μια εξολογική κρίση και κάνανε ολόκληρη σύνδεξη τύπου οι συνάδελφοι της, της Ε, και εγώ είχα πάει στην ε, Μισιόν. Τερικάμπρα, Αλμπιόλ, Εύη, ήμασταν, ε, ε, ήμασταν και εμείς εκεί. Πρέπει να μα μας δώσουν ευκαιρία και εμείς να μιλήσουμε. Κάνανε συνέντευξη στην έδρα της Γκουε. Κοιτάξτε, εγώ είμαι πρόεδρος, λέει η κυρία Βίξτρομ. Αυτό πάει να πει ότι τηρούμε τα όσα προβλέπονται. Δηλαδή, είχαμε αυτού του είδους την προφορική έκθεση από την επικεφαλής αντιπροσωπείας και μόλις υπάρξει ένα κείμενο θα συζητήσουμε μία έκθεση και όλοι τότε θα λάβουν το λόγο και θα μπορεί να γίνει ουσιαστική συζήτηση. Το θέμα ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ότι σας καίει όλους, αλλά εάν δώσω το λόγο ε, τώρα σε όλους τους θέλουν. Θα πρέπει οι αιτούντες να περιμένουν μέχρι αύριο το οποίο δεν είναι σωστό. Δεν συμφωνώ, καταχωρήστε το ότι δεν συμφωνώ με την Πρόεδρο. Δεν συμφωνεί η πολιτική μας ομάδα. Παρακαλώ αυτό να καταχωρηθεί στα πρακτικά. Now. Καλώς, καλώς λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα πάμε στο σημείο υπαρθυμών 9. Είναι η αναφορά 663, 663 του και αφορά τον νόμο 437 της Ελλάδος και αφορά τον κίνδυνο που διατρέχει το δικηγορικό λειτουργήμα εξ αυτού του νόμου. Καλωσορίσατε οι ετούντες εδώ στην Επιτροπή μας. Ζητούμε συγγνώμη για οποιοδήποτε πρόβλημα θα είχατε και που έπρεπε να το ε, ξεπεράσετε για να φτάσετε μέχρι εδώ. Οπότε έχουμε εδώ τον κύριο Γιώργιο Μπέσκο και τον κύριο Αλεξάνδρο Μανολόπουλο. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά ο καθένας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αξιότιμοι ευρωβουλευτέ και κυρία Πρόεδρο για την τιμή που μα κάνατε να παρασταθούμε ενώπιόν σας ανταποκρινόμενοι άμεσα στην αίτηση και καταγγελία που υποβάλαμε. Το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο διασφαλίζει ρητά τα δικαιώματα της ιδιοκτησίας και της περιουσίας ο Χάρτη των Δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 7 Δεκεμβρίου 2000, που αποτελεί τμήμα τη μεταρρυθμιστική συνθήκη τη Λισαβόνα, υιοθετεί ρητά την προστασία τη αξιοπρέπεια του ανθρώπου ω αξία κατά το άρθρο 1 και 2, κατά το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στι αξίε του σεβασμού τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια ω θεμελιώδη δικαίωμα. Δυστυχώ, οι ανωτέρω θεμελιώδει αρχέ που πρέπει να διέπουν την ευρωπαϊκή ε, κοινωνία δεν ισχύουν στη χώρα μας για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους δικηγόρους. Η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προχώρησαν στην ψήφιση του ασφαλιστικού και φορολογικού νόμου, νόμων, οι οποίοι συνδυαστικά μας έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο. Κυριολεκτικά αυτό που λέμε στην αναφορά μου καταγγελία μας δίμηση περιουσίας είναι αληθές. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία τα οποία αναφέρουμε, προκύπτει από τα γραμμάτια προείσπραξη, προκύπτει από τι κρατήσει και στο οποίο καταδεικνύεται ότι από το συνδυασμό των δύο αυτών νομοσχεδίων δεν υπάρχει κανένα ελπίδα, κανένα δικαίωμα ε, και καμία ε, διέξοδος για μας. Έχουμε φτάσει σε αδιέξοδο. Και το χειρότερο ποιο είναι, ότι μετά την καταγγελία μας ψηφίστηκε πρόσφατα νόμος, βάσει του οποίου αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές πλέον 16%, καθώς θεωρείται εάν είναι δυνατόν, ότι οι ασφαλιστικές δαπάνες είναι εισόδημα, οπότε ανεβαίνει ο συντελεστής βάσει του οποίου θα γίνει η παρακράτηση των εισφορών. Και, και το χειρότερο ακόμα το οποίο πρέπει να το επισημάνουμε είναι ότι σε τέσσερα χρόνια οι ασφαλιστικές εισφορές από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει περίοδος εκτόσεων βάσει του νόμου θα αυξηθούν κατά 50 με 60% περίπου. Δηλαδή φτάνουμε στο σημείο το αδιανόητο ότι ξεπερνάμε το 100%. Δυστυχώς η αξιοπρεπής επιβίωση, η ανάπτυξη και η ευημερία ενός λαού χρήζει κυρίως ισχυρής πολιτικής βούλησης. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε σε εσά, διότι θεωρούμε ότι πλέον είστε το τελευταίο ανάγχωμα σε αυτήν την καταστροφή που έχουμε υποστεί. Αυτή η πολιτική βούληση δεν πρέπει να διαμορφώνεται μόνο από αριθμού. Οφείλει να ερευνά την πραγματική οικονομική και κοινωνική διάσταση αυτών των αριθμών, να αφογκράζει τι αντοχέ μα. Γι' αυτό σήμερα βρίσκομαι ενώπιον σα ω επιστήμονα, ω ελεύθερο επαγγελματία, ω Ευρωπαίο πολίτη, πάνω απ' όλα σα ω άνθρωπο και σα δηλώνω ότι οι Έλληνε πολίτε, εμεί οι δικηγόροι, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίε, που Είμαστε ομοκλώ ανάπτυξη μια χώρα, δεν αντέχουμε να σηκώσουμε άλλο αυτό το βάρο τη οικονομική ύφεση. Έχουμε καταστραφεί. Το κράτος εφαρμόζει νόμους ληστρικής πολιτικής σε βάρος της εργασίας μας και της περιουσίας μας. Δυστυχώς, δεν έχουν καταλάβει κάποιοι ότι η μοχλός ανάπτυξη σε μια κοινωνία είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία, οι ελεύθεροι επαγγελματίε οι επιστήμονες. Από τη στιγμή που μας καταστρέφει η ελληνική κυβέρνηση στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης, δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος και γι' αυτό η χώρα μας βρίσκεται σε τόσο παραδεταμένη ύφεση θεωρούμε ότι πρέπει πλέον εσείς που εκπροσωπείτε τους Ευρωπαίους πολίτες, γιατί εσείς αφού την ιδιοσυγκρασία των λαών και τα συναισθήματα της κοινή γνώμη και τα αισθήματα, πρέπει να διαμορφώσετε με μια ισχυρή σας πολιτική παρέμβαση ένα καθεστώς το οποίο πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματά μας. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο αδιέξοδο, τα οποία νομίζουμε ότι μόνο εσείς είστε η ελπίδα μας. Πρέπει δηλαδή να πάρετε εσείς την κατάσταση στα χέρια σα μέσα από την πολιτική βούληση που έχετε, η οποία και πρέπει να είναι ισχυρή. Ε, εμείς τώρα είμαστε καταστραμμένοι ουσιαστικά, δυστυχώς. Αλλά έχουμε, οφείλουμε στις νεότερε νεότερες γενναίες, στους νεότερους δικηγόρους, στους νεότερους επαγγελματίες, να τους δώσουμε κι εμείς μια ελπίδα, μια δυνατότητα να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να εργαστούν. Αυτά που λέμε δεν είναι υπερβολικά, είναι κυριολεκτικά. Αυτά τα οποία λέμε δεν τα λέει κανείς, γιατί μέσα οι τεχνοκράτες, μέσα από κάποιες ε, διεργασίες που κάνουν, δεν μας βλέπουν ως άνθρωπους με δικαιώματα, μας βλέπουν ως αριθμούς. Θέλουμε και παρακαλούμε να μας δείτε ως άνθρωπους, γιατί εσείς εκπροσωπείτε εμάς και η ε, πολιτική σας απόφαση, κατεύθυνση πρέπει να είναι άμεση και ε, καθοριστική. Πλέον δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ούτε για αναβλητικές ε, ε, διεργασίες ούτε για τίποτα άλλο. Έχουμε καταστραφεί και πλέον δεν μπορούμε άλλο. Παρακαλούμε για την ανταπόκριση στο έτοιμά μας. Είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες και αξίζουμε το σεβασμό όλων. Ευχαριστώ. Αξιότιμα... Can I, πριν δώσω σε οποιονδήποτε το λόγο, να ζητήσω από τους συμβούλους του ΕΛΚ να κάνουν λίγο περισσότερη ησυχία και να καθίσουν. Now the floor is yours. Τώρα έχετε το λόγο. Και συμπαθάτε με. Ε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, ε, χαιρόμαστε ιδιαίτερως που βρισκόμαστε στο λίκνο της προάσπισης των δικαιωμάτων μας ως Ευρωπαίων πολιτών και κυρίως ως επιστημόνων. Συμπληρωματικό σε αυτά που ανέφερε ο κύριος Πρόεδρος, αυτό που θέλω να τονίσω και θεωρώ ότι έχει διαφανεί από το σώμα της αναφοράς μας και τα υπομνήματα και έγγραφα που έχουμε αποστείλει και έχετε όλοι στη διάθεσή σας, είναι διότι ότι δια του ασφαλιστικού και φορολογικού νόμου σορευτικός, τη σορευτικότητα των οποίων είτε λησμονεί είτε επιλησμονεί η Κομισιόν στην απάντηση που απέστειλε, θίγεται ο σκληρός απολύτως προστατευτέως πυρήνα θεμελιωδών συνταγματικών δικαιωμάτων και κυρίω θεμελιωδών δικαιωμάτων του πρόσθετου πρωτοκόλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Θίγεται η ίδια η ανθρώπινη αξία που ενυπάρχει σε κάθε δικαίωμα που προστατεύεται και προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ε, θίγεται ε, λοιπόν η αξιοπρεπής διαβίωση του πολίτη μιας χώρας που ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια, επομένως επί εσφαλμένης προϋποθέσεως, είτε απολύτως αβασίμως, κινείται ο ισχυρισμό της Κομισιόν ότι για τα τεθέντα ζητήματα αποκλειστικά αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια. Ε, είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν συνετάγησαν ασφαλιστικές ε, αναλογιστικές μελέτες, όπως ψευδώς αναφέρει στην απάντησή της η Κομισιόν για τον ασφαλιστικό νόμο, και τούτο προκύπτει αδιαφυσβήτητα και αναντήρητα από τα προσκομιστέντα εφημών έγγραφα και από το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο της χώρας μας, ή το ελεγκτικό συνέδριο. Ε, ψηφίστηκε ένα στην ουσία αμυγός πρακτικός νόμος φορολογικής υφής που εξαϊλώνει οποιοδήποτε από κερδενόμενο εισόδημα του ελεύθερου επαγγελματία, είτε μικρό είναι τούτο, ε, είτε μεγάλο. Χιλιάδε ελεύθεροι επαγγελματίε έχουν εξαναγκαστεί από τι υπέμενε επιβαρύνσει σε πάυση τη λειτουργία του επαγγέλματό του. Εμεί δεν λειτουργούμε ούτε σκεπτόμεθα με μηδενιστική βάση ω προ τον ασφαλιστικό και φορολογικό νόμο. Αυτό που ζητούμε είναι σεβασμό τη αρχή τη αναλογικότητα. Και συναστηματικά φορτισμένη λέξη σεβασμό στην αρχή αυτή που συναντάται αυτούσια μόνο στο άρθρο 2 του ειδικού μα συντάγματο αλλά και στην Ευρωπαϊκή ε, Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δηλαδή στο σεβασμό τη αξία του ανθρώπου, σημαίνει ότι η αρχή αυτή παραγνωρίζεται από τον κοινό νομοθέτη ή και ακόμα από τη δικαστική εξουσία. Αυτή την αρχή λοιπόν εσεί καλείστε να αντιθέσετε στα όρια που τη αρμόζουν, τη αυτά του απόλυτου σεβασμού, η αρχή αυτή είναι από τι βασικότερε αρχέ που πρέπει παρεγκλήτω να τηρεί και η κρατική εξουσία και η δικαστική και σε συγκεκριμένη περίπτωση θα βρει εφαρμογή με την εκλογήκευση των ποσοστών των ασφαλιστικών και φορολογικών επιβαρύσεων σε τέτοιο σημείο που θα μπορέσουν άπαντε να δυνηθούν και οι επιστήμονε δικηγόροι και οι ε, λοιποί ελεύθεροι επαγγελματίε να ανταποκριθούν στα ασφαλιστικά και φορολογικά του βάρη και τι εν γέννη υποχρεώσει του όχι δημοβωμένου όμω του εισοδήματό του και καταπαραθρούμενη τη αξιοπρέπεια και τη αξιοπρεπού διαβίωση αυτών και των οικογενειών του. Και ναι, μεν μπορεί κάποιο να σκεφτεί ότι η χώρα μα διέρχεται μια σοβαρή οικοδομική κρίση, όντων όμω ημών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των αξιών και οραμάτων από τι οποίε αυτή εμφορείται, ο άνθρωπο και κυρίω τα μέλη του συλλόγου που εμεί εκπροσωπούμε του επιστημονικού δεν πρέπει ποτέ να ακολουθούν σε σπουδαιότητα την όποια αναγκαιότητα δημοσιονομικής προσαρμογής. Γιατί το κράτος είναι πρωτίστως οι πολίτες του και σήμερα καλείστε να αποδείξετε κατά πόσον οι αξίες στις οποίες θεμελιώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αξίες κατ' όνομα, αλλά αξίες εν της πράγμαση προστατευόμενες και αναγνωριζόμενες από εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίνω τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Λάινε, ο κύριος Καρόνε. Θα μοιραστείτε τον λόγο. Μιλάει ο κύριος Λάινε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα οι κανόνες εναρμόνισης εισπορών οριστήκαν στο νόμο 4387 του 16 το λεγόμενο συνταξιοδοτικό νόμο στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του, συνταγμα... του συνταξιοδοτικού συστήματος για την επίτευξη της βιωσιμότητάς του καθώς στα πλαίσια του οικονομικού προγράμματος χρειαζόταν εξοικονόμηση εξόδων. Ένας στόχος της μεταρρύθμισης είναι η σύνδεση μεταξύ ωφελών και εισφορών. το οποίο επιτυγχάνει βάζοντας τους αυτοαπασχολούμενους στην ίδια κατηγορία όπως άλλους εργαζόμενους καθώς υπήρχαν εισπορές που βασίζονταν σε ένα τεκμαρτό εισόδημα τα χρόνια άσκησης ενός επαγγέλματος αυτό άλλαξε τώρα πλέον βασίζονται στο φορολογητέο εισόδημα κατά το τελευταίο φορολογικό έτος. Οπότε είναι στα, πλαίσια, στα ίδια πλαίσια όπως άλλες κατηγορίες εργαζόμενων. Παρά τα αυτά υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις για την προστασία από απότομες αλλαγές έως το 2020 Υπάρχει μια μεταβατική περίοδος για την αύξηση των εισφορών. Υπάρχει επίσης μια εξαίρεση για νέους εργαζόμενους, οι οποίοι επί τέσσερα χρόνια μπορεί να έχουν χαμηλότερες εισφορές όσον αφορά την οικονομική μελέτη που αναφέρθηκε στην παρέμβαση ενός των αναφερόντων αυτή συνόδευσε τον συνταξιδοτικό νόμο ήταν πολύ λεπτομερής και περιεκτική και σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές διασφάλισε τη χρήση όλων των παραμέτρων στη μελέτη αυτή έτσι ώστε να μπορεί να διασφαλιστεί η νομιμότητα της μεταρρύθμισης. Πέραν αυτού, Πιστεύω πως αυτά είναι τα κυρίως ζητήματα που ήθελα να θέσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα ανοίγω τη συζήτηση του κ. Ζαριανόπουλος πρώτος. Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας ότι μετά από την κατάσταση της αναφοράς έχουμε και εξελίξεις. Η... Το ασφαλιστικό στην Ελλάδα με το τέταρτο μνημόνιο που υπέγραψε η σημερινή κυβέρνηση έχει γίνει πολύ χειρότερο από αυτά που ακούσατε. Αναφέρθηκε και από τον ε, ε, εκπρόσωπο εδώ των αναφερομένων ότι ένα από τα τελευταία μέτρα που έχει υιοθετηθεί στη χώρα μας είναι να φορολογηθούν ακόμα και οι ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή περιουσία η οποία δεν υπάρχει. Ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να τονίσουμε είναι βεβαίως θίγονται οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, θίγονται βεβαίως όμως και όλες οι υπόλοιπες ε, ομάδες των αυτοαπασχολούμενων, θίγονται οι εργαζόμενοι, θίγονται οι συνταξιούχοι με τρομακτικές για 16 φορές περικοπές των συντάξεων και βεβαίως οι νέοι εργαζόμενοι. Η απάντηση που δόθηκε από την Κομισιόν στην αναφορά είναι κυριολεκτικά προκλητική. Ποιος δεν γνωρίζει ότι η Κομισιόν προσυπογράφει τα κείμενα των μνημονίων που με μεγάλη λεπτομέρεια αναφέρονται στην υποχρέωση να μειωθούν οι συντάξεις, να αυξηθούν οι εισφορές, να τσακιστεί η κοινωνική ασφάλιση. Είναι ψεύτικη η απάντησή της και μάλιστα όταν έχει, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε όλα τα μνημόνια και συνεχίζει στην κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης. Γιατί άλλωστε το διακηρύσει δημόσια. Στα κείμενά της για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, τα επανειλημμένα κείμενά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει στη μεταρρύθμιση των διεξοδικών συστημάτων, ώστε να γίνουν φιλικά στην ανάπτυξη. Με λίγα λόγια, να μην εισφέρουν οι εργοδότες, να μην υποβοηθά το κράτο το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης και ό,τι εξοικονομείται από το κράτος από αυτήν την περικοπή να δίνεται σε μεγάλες επιχειρήσεις ως κίνητρο για την κερδοφορία τους. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στο ίδιο νομοθέτημα πρόσφατο, το τέλο του μνημονίου, με το οποίο αυξάνεται η φορολογία ακόμη και των πιο φτωχών αυτών που ε, βγάζουν ένα εισόδημα της τάξης των 300-400 ευρώ το μήνα, στο ίδιο νομοθέτημα μειώνεται η φορολογία των μεγάλων επιχειρήσεων κατά 3% προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως και οι ελληνικές κυβερνήσεις που συνεργάζονται μαζί της, να κατεδαφίσουν την κοινωνική ασφάλιση και να την αντικαταστήσουν με την ιδιωτική ασφάλιση και με τα επαγγελματικά ταμεία. Ένα νέο πεδίο κερδοφορία. Ορισμένα στοιχεία που αναφέρονται στην έκθεση νομίζω ότι είναι καλό να ακουστούν στην αναφορά, με συγχωρείτε, να ακουστούν και εδώ για να καταλάβει ο καθένα την έκταση τη φαγή. Για του αυτοαπασχολούμενου μιλάμε και για του δικηγόρου. Με το νομοθέτημα στο οποίο αναφέρεται η, η αναφορά θα επιβάλλεται, επιβάλλεται μάλλον εισφορά για την κύρια σύνταξη 20% επί του εισοδήματος. Εισφορά για την επικουρική σύνταξη 7,5% επί του εισοδήματος. Εισφορά για την υγεία περίπου 7% και εισφορά για το εφάπαξ 4%. Αυτό μας κάνει 38,5% ασφαλιστικές εισφορές επί του εισοδήματος. Και αν προσθέσουμε 26% φόρο πηγαίνουμε στο 64,5% ασφαλιστική και φορολογική επιβάρηση. Και δεν σταματάμε εδώ. Άλλο 26% φορολογική επιβάρηση για την προκαταβολή του φόρου του επόμενου έτους. Καταλαβαίνετε ότι δεν απομένει τίποτα. Ακόμα και στο μηδενικό εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων πρέπει να πληρωθεί φόρος 2.700 ευρώ σε ανύπαρκτο εισόδημα. Έτσι ξεκινάνε οι κατασχέσεις και οι πληστεριασμοί απέναντι σε χιλιάδε εντό εισαγωγικών οφειλέτες του δημοσίου που εξελίσσονται. Στην πραγματικότητα και για το συγκεκριμένο επάγγελμα τι κάνει αυτό ο νόμο, όπω και για τι υπόλοιπε ομάδε των αυτοαπασχολούμενων. Πετάει κυριολεκτικά έξω από το επάγγελμα του νέου, του φτωχότερου δικηγόρου και του άλλου αυτοαπασχολούμενου για να ενισχυθούν τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία, οι μεγάλε νομικέ εταιρείε, όπω και οι μεγάλοι του κάθε κλάδου. Αφήστε δε για το ποια σύνταξη μιλάμε. Γιατί ύψο σύνταξη και με ποιε όρου. Στα 40 χρόνια δουλειά και βεβαίω με μια εθνική σύνταξη βασική 384 ευρώ και μετά ό,τι σου αναλογεί, ανάλογα βέβαια και με τα μειωμένα εισοδήματα και τις μειωμένες φορές σου και τις, τα μειωμένα εισοδήματα σε όλη τη διάρκεια τη επαγγελματική σου ζωή. Συμφωνώ με την ουσία της αναφοράς. Απόλυτα. Έτσι είναι η κατάσταση. Αλλά διαφωνώ με έναν ε, χαρακτηρισμό. Είναι πολιτική η διαφορά, μην την, ε, δεν είναι κάτι άλλο καμία ελπίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σφαγείο είναι και σφαγείο θα συνεχίσει να είναι. Η παρέμβασή μα εδώ έχει την έννοια και να αναδείξουμε το ζήτημα και να πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Εμεί, σαν κουκουέ δεν έχουμε καμιά ελπίδα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο επιμένουμε παρά την προκλητική ε, απάντηση τη ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η αναφορά να μείνει ανοιχτή και να συνεχιστεί η περαιτέρω διαρρεύνηση και με τα νέα στοιχεία που έχουν εισφερθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τους αναφέροντες οι οποίοι έφεραν το ζήτημα αυτό στην ε, Επιτροπή μας. Πήραν μια πρωτοβουλία ουσιαστικά εκπροσωπώντας όχι μόνο τον Σύλλογο, Δικηγορικό Σύλλογο του Αιγείου, αλλά επί της ουσίας εκπροσωπούν πλέον όλο τον δικηγορικό κλάδο της Ελλάδος. Και στην πράξη εκπροσωπούν τους ελεύθερους επαγγελματίες διότι τα μνημονιακά μέτρα που έχουν επιβληθεί, που διαλύουν πλέον τους μικρομεσαίους, έχουν τον ίδιο πυρήνα. Δηλαδή ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο επί της ουσίας επιβάλλει τεράστιες ασφαλιστικές εισφορές, μία φορομπηχτική πολιτική η οποία οδηγεί σε φορολοηλασία. Επομένως η αναφορά αυτή είναι πολύ τυπική του τι συμβαίνει στην Ελλάδα μια κατάσταση που έχει επιδεινωθεί με το τέταρτο μνημόνιο, με επιπλέον σκληρά μέτρα και όλα αυτά υποτίθεται για να υπήρχε ρύθμιση του χρέους που όπως είδαμε στο τελευταίο Eurogroup δεν έγινε. Δεύτερο, να ευχαριστήσω την Επιτροπή μας η οποία αποδέχτηκε το δικό μου αίτημα να εξετάσουμε με την κατεπίγουσα διαδικασία αυτή την αναφορά διότι πράγματι τα ζητήματα επίγουν και νομίζω ότι η ανάλυση από πλευράς των αναφερόντων έχει καταδείξει το ζήτημα αυτό. Τρίτο, θα πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η θέση της Κομισιόν όχι μόνο επί της ουσίας τι είπε, θα αναφερθώ σε αυτά, αλλά ποιος είναι ο ρόλος της. Και είναι κάτι που το είπα και στον κύριο Τίμερμανς όταν είχε έρθει στην Επιτροπή μας, στον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, ότι όταν ε, λαμβάνει μια αναφορά η Κομισιόν, δεν πρέπει απλά να ρωτάει το κράτος μέλος και να παπαγαλίζει τις απόψεις που λέει κάθε κράτος, <laughs> γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Η Κομισιόν πρέπει να μπει σε βάθος, να ρωτήσει, να αμφισβητήσει, να δει τι γίνεται. Διότι αυτά που μας είπε η Κομισιόν επί τη ουσία, είναι αυτά που ισχυρίζεται και η ελληνική κυβέρνηση. Δεν εξέτασε την υπόθεση σε βάθος. Και θα σας πω γιατί δεν το έκανε. Διότι υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων, το έχουμε ξαναπεί. Η Κομισιόν από τη μια υποτίθεται ότι υπερασπίζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δίκαιο συνολικά των πολιτών και από την άλλη στην περίπτωση της Ελλάδας είναι μέλος της Τρόικας, έχει συμφωνήσει με αυτά τα μέτρα και έχει επιβάλει ουσιαστικά μαζί με την ελληνική κυβέρνηση αυτά τα μέτρα. Άρα τι θα υποστηρίξει η Κομισιόν. Θα υποστηρίξει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δίκαιο των αναφερόντων ή θα υποστηρίξει τις απόψεις της ίδιας της Τρόικας. Εκεί βρίσκεται η υπόθεση. Ερχόμαστε τώρα επί της ουσίας. Νομίζω ότι αναφέρθηκε ξεκάθαρα ποιο είναι το ζήτημα. Πρώτον, πλήττεται το δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση. Δεύτερον, πλήττεται το δικαίωμα στο, στην άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος, διότι με αυτούς τους όρους, όταν ουσιαστικά το 80% του εισοδήματος που θα εισπράξει κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας, δικηγόρος στο Αίγυο, θα πάει στο κράτος, το απομένει μόνο 20% να συντηρήσει το γραφείο του, να ζήσει, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Και τρίτον, πλήττεται το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, διότι πάλι του αφαιρούνται τα περιουσιακά δικαιώματα και οδηγείται σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει μέλλον πλήττεται η αρχή της αναλογικότητας που υποτίθεται ότι υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε παραβίαση δικαιωμάτων τα οποία προστατεύονται, I'm going to finish, τα οποία προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού? Από τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Άρα εδώ θα περίμενα από την Κομισιόν να πει ότι εξετάζει το θέμα, ότι προχωρεί παραπέρα και ετοιμάζεται να παραπέμψει την κυβέρνηση, την χώρα, διότι εν προκειμένου παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραβιάζει τα δικαιώματα των αναφερόντων. Άρα λοιπόν η πρότασή μου κυρία Πρόεδρε συγκεκριμένη. Πρώτον, η αναφορά θα πρέπει να μείνει ανοιχτή. Δεύτερον, να στείλουμε επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να δώσουν εξηγήσει για ποιο λόγο παραβιάζουν εν προκειμένου τα δικαιώματα των αναφερόντων όπως αυτά προστατεύονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτον, να ενημερώσουμε και να ζητήσουμε την γνώμη της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής εδώ του δικού μας Κοινοβουλίου, όπου εκεί υπάρχει ένα working group που ασχολείται με τα θέματα του μνημονίου στην Ελλάδα. Γιατί αυτό είναι σοβαρό ζήτημα. Και επίση πιστεύω ότι και η Επιτροπή ε, του Κοινοβουλίου μας που ασχολείται με τα εργασιακά θα πρέπει να λάβει υπόψη της τι συμβαίνει. Άρα λοιπόν αυτές είναι οι προτάσεις μας να ληφθούν υπόψη και φυσικά αφού ακούσουμε και τους συναδέλφους να καταλήξουμε σε μια απόφαση την οποία βεβαίως εσείς θα μας προτείνετε για να προχωρήσουμε παραπέρα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ και τώρα θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο σύντομοι γιατί έχουμε για 15 λεπτά ακόμα τους διερμηνεί. Έχουμε ακόμα δύο ομιλητέ. Παρακαλώ να είστε σύντομοι και μετά θα δώσουμε το λόγο πάλι στους αναφέροντες. Ο κ. Ευχαριστώ πρόεδρε και θα είμαι σύντομο. Η οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα είναι δραματική. Δεν γνωρίζω ακριβώ τι σημαίνει η νέα νομοθεσία, αλλά πολύ φοβάμαι ότι είμαστε σε πειρασμό να ζητάμε από την Ελλάδα και από τους φορολογούμενους αυτά που ζητάμε από τους Δανούς και τους Γάλλους. Θα πρέπει να επανεξετάσουμε την κατάσταση λοιπόν εκεί. Σύμφωνα και βάσει των δραματικών συνθήκων που έχουν. Οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται χρόνο και συμφωνία από το λαό προκειμένου να υποστηριχθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό ζητώ από την ομάδα να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Όπως είπε και ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ. Εξαιρετικά. Ο κύριος Γιάρ. Ναι, Να ξεκινήσω με το συμπέρασμα. Θα ήθελα και εγώ να μείνει ανοιχτή η αναφορά, αλλά με μια, για ένα άλλο λόγο από αυτό που ανέφερε ο Κύριος Μαριάς. Θα ήθελα να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ξέρω πώς γίνεται ένας ε, μέσος ε, εισοδηματίας να πρέπει να δίνει 80% του εισοδηματός του. Είναι αποθαρρυντικό. Σε ό,τι αφορά δηλαδή το να πληρώνει 80% των εισοδημάτων του. Θέλω να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Για να ρωτήσω, όντως ισχύει κάτι τέτοιο γιατί η πρόθεση της οικονομίας και των μικρομεσαίων είναι διαφορετικό πράγμα. Με διαφορετικό τρόπο διαμορφώνεται. Θα πρέπει να τους υποστηρίξουμε και είμαι... Έχω την εντύπωση ότι κάποιες περιπτώσεις οι προτάσεις ε, της κυβέρνησης δεν είναι αποτεκτές. Και μετά ρίχνει το φταίξιμο στις Βρυξέλλες. Ε. Α, ότι οι Βρυξέλλες θέλουν να κάνουμε οικονομίες. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμα πολλά χρήματα σε μαύρους λογαριασμούς, τα οποία δεν τα πειράζει κανείς. Και νομίζω ότι χρειάζεται μεγάλη ε, συνένεση από τον κόσμο. Θα πρέπει να γίνουν τα πράγματα αυτά με δικαιοσύνη. Να υπάρχει ε, η αίσθηση της δικαιοσύνης. Να παραμείνει ανοιχτή λοιπόν και να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει κατά πόσον όντως ισχύουν αυτά. Εγώ είμαι από την Ανατολική Γερμανία και τότε οι μικρομεσαίοι φορολογούνταν 90%. Ήταν κλασικό σημάδι αυτό του κομμουνισμού. Δεν πειράζει, θα δώσουμε όλα στο κράτος. Μα δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν έτσι τα πράγματα, γιατί de facto αυτά δεν μπορούν να ισχύουν. Αν ισχύουν όλα αυτά, πραγματικά ε, πρέπει να το κοιτάξουμε. Να μην είναι λοιπόν ανοιχτή η αναφορά και να τσεκάρουμε κατά πόσο ισχύουν πραγματικά όλα αυτά. Κύριε Πρόεδρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι ολοκληρώνω το κατάλογο των ομιλητών, των συναδέλφων και να δώσω το λόγο πάλι σε εσά για δύο λεπτά στον καθένα. Κυρία Πρόεδρε, <clears throat> πραγματικά στενοχωρήθηκα από την τοποθέτηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι πλέον δείχνει ότι ο ρόλο τη δεν είναι αυτό που πρέπει να έχει βάσει τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τη Ευρωπαϊκή θέση που πρέπει να έχει. Είναι απαράδεκτο να έρχεται εδώ και να λέει ψέματα. Γιατί έχετε και διαψεύδει η ίδια το ανώτατο δικαστήριο της χώρας μας, το οποίο είπε ότι δεν υπάρχει αναλογιστική μελέτη. Όταν, τα Όταν το κατατεθένομο σχέδιο ε, κατατέθηκε στη Βουλή χωρί αναλογιστική μελέτη και η μόνη αναλογιστική εντό εισαγωγικών, ούτε εντό εισαγωγικών, γιατί δεν είναι μελέτη, ένα ενημερωτικό σημείωμα ήταν, το οποίο καταδεικνύει αυτό το πράγμα. Εγώ στεναχωριέμαι και πραγματικά μου κάνει εντύπωση ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δείχνει ότι δεν είναι αυτό ο ρόλο που πρέπει και έχει και έχω απέτηση και εγώ σαν Ευρωπαίο πολίτη να κοιτάξει την καταγγελία μα, να δει γιατί υποφέρουμε και, και δεν μπορούμε να ζήσουμε και κάθεται τώρα μαζί με την ελληνική κυβέρνηση όπω συντάσσουν του νόμου αυτού σε συνεργασία και παίρνει τι τοποθετήσει τη ελληνική κυβέρνηση. Αυτό είναι απαράδεικτο και δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο, δεν, συνάδει με τον ευρωπαϊκό χάρτη, με, μια Ευρώπη που ονειρευόμαστε όλοι. Γιατί η Κομισιόν, όπω τα λέει αυτά τα πράγματα, προφανώ δεν αδιαφορεί για την ανθρώπινη διάσταση όλων μα. Ε, κοιτάνε μόνο να μα βλέπουν σαν αριθμού, δεν δίνουν καμία ε, σημασία στην αξία και στην αξιοπρεπιά μα, στο δικαίωμα τη επιβίωσή μα, στο δικαίωμα τη ζωή μα. Και όλα αυτά που λέει και ουσιαστικά η ίδια ότι έχουν δώσει τέσσερα χρόνια μεταβατικό διάστημα. Ε, λοιπόν, αυτά τα τέσσερα χρόνια δεν είναι μεταβατικό διάστημα, γιατί μετά την πάροδο των τεσσάρων ετών, το 80% που υπάρχει τώρα σε δίμευση θα γίνει 140% γιατί θα φύγουν αυτέ οι εκτόσει. Και το χειρότερο και γι' αυτό δεν αναφέρει και τίποτα γι' αυτό, εμεί κάναμε καταγγελία σε συνδυασμό με το φορολογικό και το ασφαλιστικό. Για το φορολογικό τίποτα. Έτσι. Αυτό καταδεικνύει λοιπόν ότι δεν έχει να πει κάτι και πρέπει επομένω και εσεί, σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να δώσετε στην Κομισιόν να καταλάβει ότι πρέπει να λειτουργεί για το συμφέρον του Ευρωπαίου πολίτη, του Ευρωπαίου άνθρωπου και όχι τεχνοκρατικών και οικονομικών συμφερόντων που δεν συνάδουν με το ευρωπαϊκό όραμα. Ευχαριστώ πολύ. Συμπληρωματικό, ε, και μόνο κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τους ε, κυρίους ε, Ευρωβουλευτές. πραγματικά στόκευσαν και κατάλαβαν ακριβώς ποιο είναι το ζήτημα που απασχολεί τον κλάδο μα και τους λοιπού ελεύθερου επαγγελματίες. ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μαριά και τον κύριο Σαριανόπουλο. Πραγματικά εξέτασαν, τα, έχουν δει τα στοιχεία του φακέλου, φάνηκε από τις απαντήσεις τους. Και καταλήγοντας να κάνω μια μικρή μόνο παρατήρηση, ε, με την καλή έννοια πάντα, ε, στον κύριο βουλευτή εξ Ανατολικής ε, Γερμανίας, ο οποίος είπε να κοιτάξουμε αν είναι ε, πραγματικά το ποσοστό της επιβαρύνσεως στο 80%. Ε, θέλω να σας αναφέρω ότι είναι αισιόδοξε αυτές οι προβλέψεις. Η επιβάρυνση είναι πολύ μεγαλύτερη εμείς ε, αποτινόμαστε σε εσάς, ελπίζουμε σε εσάς. πραγματικά πρέπει να ληφθούν οι δράσεις τουλάχιστον στο πλαίσιο που ανέφερε ο αξιότιμος βουλευτής Ευρωβουλευτής, ο κύριος ε, Μαριάς. Ευχαριστώ πολύ. Yes, thank you very much. And... Uh, ναι, ευχαριστώ πολύ και τώρα έφτασε η ώρα να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα σχετικά με αυτήν την αναφορά. συνάδελφοι πρότειναν να παραμείνει ανοιχτή για πολλούς λόγους και να επανέλθουμε στην Επιτροπή. Και αυτό που θα ήθελα να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μας είναι να αξιολογήσει πιο πολύ εις βάθος το έγγραφο που μόλις χτες απεστάλλει από τον Έλληνα Υπουργό Εργασία και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το οποίο ονομάζεται έγγραφο τοποθέτησης. Το λάβαμε μόλις χτες, σας το προωθήσαμε στο έγγραφο αυτό γράφουν πως οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης συνδέονται πλέον με το πραγματικό εισόδημα και όχι ένα τεκμαρτό εισόδημα πλέον. Και θα ήθελα, θα ήθελα να μάθω αν αυτό ισχύει ή όχι. Και έχουμε εμπιστοσύνη στην Επιτροπή η οποία θα το κοιτάξει και θα μας φέρει περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες γι' αυτό. Επίσης θα θέλαμε να εργαστεί λίγο περισσότερο επί του πλαισίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίως τι έγινε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 18 Μαΐου μετά από μια αποκαταρκτική συμφωνία στο πλαίσιο του Euro Working Group. Πρέπει να τα εξτάσουμε επίσης. Επίσης, μπορούμε να, πρέπει να πεταθούμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και επίσης τον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφαλείας για να εκφράσουμε την ανησυχία μας για το ζήτημα. Πιστεύω πως θα πρέπει να επανέλθουμε μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας να ζητήσουμε τον Έλληνα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουν ένα έγγραφο τοποθέτηση, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν έχουν μια βιώσιμη λύση ή ένα, ή ένα συμβιβασμό για την επίλυση του προβλήματος αυτού. Υπάρχει μόνο μια τοποθέτηση. Ίσως θα πρέπει να, ρωτήσουμε, να ζητήσουμε κάτι περισσότερο από αυτούς όσον αφορά τις πληροφορίες. Κύριε Μαραριά, έχετε να πείτε κάτι. Στο ότι πρέπει να απευθύνουμε, ε, I'm going to, to say it again for Peter, ε, συμφωνώ με την πρότασή σας ότι πρέπει να απευθύνουμε επιστολή και στο Υπουργείο Οικονομικών και όπως είπατε και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ζητώντας τις εξηγήσει πώς πρόκειται να αντιμετωπίσουν το αίτημα και την αναφορά των αναφερόντων. Όχι να μας στείλουν ένα χαρτί γενικώ που λέει αριθμούς. Εδώ έχουμε μία αναφορά η οποία βάζει τα ζητήματα. Οφείλουν να απαντήσουν συγκεκριμένα. Επομένως στις προτάσεις σας όλες αυτές συμφωνώ όπως επίσης και να απευθυνθούμε και στον ESM όπως είπατε και στα υπόλοιπα όργανα αλλά να υπάρχει έγγραφο δικό μας απευθείας στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ζητώντας εξηγήσει και αναφέροντας ε, our concerns, τις, ε, τους, ε, τις ανησυχίες μας για το τι συμβαίνει και ζητώντας εξηγήσει. Και νομίζω ότι αυτό είναι κρίσιμο και συντόμως ελπίζουμε να απαντήσει η ελληνική κυβέρνηση για να ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα το κάνω με όλα αυτά δεν έχουμε μόνο αναφορές, έχουμε άνθρωποι εδώ μαζί μας σήμερα. Και γι' αυτό θα το κάνουμε όλα αυτά, ε, συμφωνούμε όλοι. Σας ευχαριστώ για σήμερα και, και καλή, καλή, καλό ταξίδι πολύ. πίσω στην Ελλάδα. Ευελπιστούμε σε εσάς μόνο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο να ευελπιστούμε δυστυχώς. And to all of your all colleagues, have a very nice evening and uh, see. Αποχαιρετά τους υπολείπους συναδέλφους Πρόεδρος. Καλό βράδυ.